Okay, take your seats everybody. I think we've... Uh, Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Most groups represented. Ελπίζω να εκπροσωπούνται οι περισσότερες πολιτικές ομάδες. Okay, who wanted to be here. Ε, η Βίκη και ε, και θα θέλω να είναι σήμερα εδώ, αλλά έχει συνέδριο το κόμμα τους, γι' αυτό μίλησε χθε πρώτη Βίκη. Ε, στα σημεία 7 και 8 της ημερήσιας ε, διάταξης, που είναι η οδηγία για τις ε, κεφαλαικές απαιτήσει. Ε, συνεχίζουμε την ανταλλαγή απόψεων που αρχίσαμε στο Στρασβούργο, αν θυμάστε. ο εισηγητής ο Ούντο Μπούλμαν από τους σοσιαλιστές και η Βίκη Φόρτ από τους συντηρητικούς έχουν ήδη μιλήσει, οπότε θα αναγκαστώ να μιλήσω εγώ ως κοιόδης εισηγήτρια των φιλελευθέρων και μετά ο Φιλίπ Λαμπέρς και με τη σειρά οι υπόλοιποι. Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσετε να ζητήσετε το λόγο. Και ο Γκούνα. Και ο Διέγκο Φέο. Right, so, um... Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, από τα όσα σας είπα εχθές, Washington. πρόσφατα μετέβη στην Ουάσιγκτον και νομίζω καλό θα ήταν να πούμε κάτι για τη συνολική εικόνα εφαρμογής για τη Βασιλεία 3. Ξέρουμε ότι ορισμένε χώρες θα την εφαρμόσουν νωρίτερα, ας πούμε ο Καναδάς, ε, θα έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή νωρίτερα στη μεταβατική περίοδο. Ε, αλλού οι αγορές επίσης επιβάλλουν τη ταχύτερη συμμόρφωση από ότι ε, θα επέβαλε η νομοθεσία. Δεν είναι πρόβλημα αυτό έτσι κι αλλιώς. ούτε η αντιστοιχεία βέβαια έχει πολλές ορισμούς ε, στα κείμενα που μας απασχολούν και αυτό είναι πάντα επίμαχο. Εγώ θεωρώ ότι ε, συγκρίσιμα καθεστώτα που αξίζουν αναγνώριση δεν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο αυστηρά όπως το δικό μας παντού. Μπορούν να είναι ε, αυστηρότερα κάπου αλλού και λίγο πιο χαλαρά σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις, αλλά γενικά να υπάρχει μια ισορροπία και ε, η αρμόδια αρχή ε, θα μπορέσει να αναλύσει και να βγάλει κάποια άκρη. Οι ε, ενδεχόμενε αποκλήσει Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων μπορεί να προέρθουν από την έγκριση μοντέλων ρίσκου ή κινδύνου και η εναρμόνιση που εμείς επιζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ξυλωθεί από κάποιες διαφορές στην εκτίμηση κινδύνου και η EBA θα πρέπει να μας δώσει έτσι ένα εξωτερικό καλούπι για να αναλύουμε αυτά τα μοντέλα. Και αν δούμε την ε, φερεγγιότητα 2, όπου ε, αυτή η ιδέα με τα μοντέλα ήταν καινούρια, ε, λύσαμε το πρόβλημα, αν μπορώ να πω ότι το λύσαμε, με διάφορα παράλληλα ε, μοντέλα, πρότυπα, για να δούμε τι ε, συμβαίνει με τα εσωτερικά μοντέλα. Δεν ξέρω και κατά πόσο η ε, εξέταση αυτή οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί είναι τεράστιες οι αποκλήσεις και οι διαφορές. Πάντως, αποδεικνύει αυτό που λέμε στο Κοινοβούλιο και είναι πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου, ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εξωτερικός γνώμονας για να μετρούμε ε, αυτά τα θέματα κινδύνου. Και μια ε, που μιλούμε για διεθνεί συγκρίσει, είναι και το μοντέλο του IFRS και αυτά που συζητήσαμε χτες για τα γενικά λογιστικά πρότυπα και μπορεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σας πούν τι πικρή εμπειρία έχουν από αυτές τις διαφορές που εμφανίζουν και διαφορετικά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει πάντες τώρα Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Βασιλεία και όλοι οι αρμόδιοι μελετούν αυτές τις διαφορές κυρίως στην εφαρμογή της Βασιλείας στην Αμερική και στην Ευρώπη και νομίζω είναι καλή ιδέα. Σε ό,τι αφορά ε, τώρα και το άλλο θέμα της ρευστότητας και της προοδού είναι ανοιχτά προς εξέταση, αλλά θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για την Ευρωπαϊκή ε- Ένωση και αλλού. Ε, κάτι άλλο, ε, το μηδενικό σκίνδυνο στα κρατικά ομόλογα, ας πούμε τα ελληνικά και τα γερμανικά να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο γιατί έχουν απλώς το ίδιο νόμισμα. Πρόσφατα στη Βασιλεία ε, εξετάστηκε το φαινόμενο αυτό ότι θα πρέπει να δούμε ε, το μηδενικό κίνδυνο γενικά, αλλά όταν έχουμε νομισματική ένωση ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση, τις διαφορές, θα προσπαθήσουν να το εξετάσουμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα δίκτυο, με ένα δίκτυο συγγνώμη, κινδύνου ανάλογα με τα spread και ε, να δούμε ας πούμε, ποια δημόσια κρατικά δάνεια είναι ε, καλύτερα εντό εισαγωγικών και ποια χειρότερα. Βέβαια όλα είναι σήμερα σε προκυκλική φάση, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τις κεφαλαϊκές απαιτήσει στο μέλλον. Και θα πρέπει κάποια λύση ε, να δρομολογηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον ή να ενσωματωθεί σιγά σιγά. Ένα άλλο θέμα που συνδέεται με τα δάνεια είναι η ρευστότητα και πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται τα κρατικά ομόλογα για αυτή. Δεν θα πρέπει να χαθεί πολύ κυριαρχία. Επίσης, θα πρέπει ε, βέβαια ε, τα ομόλογα να ε, θεωρούνται ως ρευστά, αλλά κάπου να υπάρχει μια τυποποίηση ε, της ποιότητας και οπωσδήποτε της διαφάνειας. Άλλο θέμα. Τα λεγόμενα buffers, μαξιλαράκια, τα αντικυκλικά πολύ συχνά ε, περιγράφονται αρνητικά. Σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καλώς, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει, μάλλον να το πω αλλιώς, εφόσον δεν υπάρχει ε, και κίνδυνο στην τράπεζα. Δηλαδή, Τώρα κανείς δεν θα τα πρότεινε αυτά. Θα ήταν ενδεχομένω ε, σκόπιμο να γίνει σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών για να ελεγχθούν οι φούσκες ε, στο ενεργητικό τους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι όμως να ελεγχθούν αυτοί και σε σχέση με την αξιολόγηση του κινδύνου και αυτό θα άξει τον ε, κόπο να ελεγχθεί <laughs> πιο στοχευμένα ε, ως άλλη μορφή ε, χρηστής μακροοικονομικής ε, διαχείρισης. Επίσης, κάποιες χώρες που έχουν μεγάλες τράπεζες με κεφάλαια πολλαπλάσια του ΑΕΠ τους έχουν αντιμετωπιστεί ή μπορούν να αντιμετωπιστούν σε κάποια ε, συστήματα, αλλά όταν ε, δεν είναι μεγάλε οι τράπεζε, είναι clusters, μπορεί να χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο buffer, μαξιλαράκι, μαξιλάρι ε, αλλά δεν μπορούμε προληπτικά να το ορίσουμε ε, ακριβώς με αυτόν τον αντικυκλικό τρόπο. Μικρές προσαρμογές στην οδηγία μπορούν να λειτουργήσουν και να εσωματωθούν και εγώ υποπτεύουμε ότι αυτό το θέμα των buffers θα μας απασχολήσει στο μέλλον και η Ευρωπαϊκή Αρχή θα πρέπει να εξετάσει τη σκοπιμότητά τους και πρόσφατα μίλησε ο Ανδρέα Αρία, ε, επανειλημμένα αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και Νομίζω το περιγράφει πολύ καλά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν κάποια διακριτική ευχαίρεια, αλλά κάπου να ελέγχεται αυτή ε, και να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει ε, κάποιος προφανής λόγος, κάποια σκοτειμότητα και όχι απλώς για να σπάσει την ανταγωνιστικότητα ή για να έχουμε προστατευτικά μέσα. Ε, υπάρχει και το θέμα ε, των τελικών χρηστών ε, στην ε, οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις και αλλού. Ελπίζουμε στο Κοινοβούλιο να έχουμε συνεπή στάση. Ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας το κείμενο, που φαίνεται ότι δεν είναι σημερινό, όταν τα ε, εργαλεία του επίπεδου 1, τα κεφαλιακά, ε, θα πρέπει να εκτιμώνται και να αποπληρώνουν. Αυτό έχει να κάνει με την εκαθάριση του πιστοτικού ιδρύματος ε, ή αφορά την επαναγορά. Δεν έχω καταλάβει καλά, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένω θα πρέπει να υπάρχει μια αρμόδια αρχή. Θα το κοιτάξουμε για την επίλυση των κρίσεων, αλλά κάπου θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις διακανονισμού που δεν είναι πλήρης εξαγορά ούτε πλήρης εκαθάριση αλλά κάποια ενδιάμεση μορφή ελέγχου ε, χαμηλών ε, κεφαλαιακών ε, δυνατοτήτων ενός πιστοτικού ιδρύματος. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ νομικίστικο, αλλά πρόσφατα μου έκανε εντύπωση αυτό διαβάζοντας για την τραπεζική επίλυση ε, σας το προτείνω λοιπόν ως ιδέα να το σκεφτείτε στις περιόδους κρίσεων ε, πριν λήξει η προθεσμία ε, των τροπολογιών. Έχω πάρα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά σταματήσω εδώ και να πάει το λόγο ο Φιλίπ Λάμπερς. So get... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάρων. Πριν περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες θα ήθελα να υπογραμμίσω τους στόχους τους οποίους θα θέλαμε η οδηγία αυτή να στοχεύσει. Καταρχάς βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου Κατά βάση οι άνθρωποι πρέπει να εξυπηρετήσουν την οικονομία και η οικονομία πρέπει να εξυπηρετήσει την χρηματοπιστωτική λειτουργία. Βασικός στόχος της οικονομίας της αγοράς στην παρούσα φάση είναι να διασφαλίσει ότι η χρηματοπιστωτική βιομηχανία αποδίδει και οδηγεί σε πάρα πολλά κέρδη. Εμείς πιστεύουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρός, αλλά θα πρέπει να υπηρετεί την οικονομία και όχι αντίθετα. Δεύτερος στόχος τον οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε και συνδέεται φυσικά και με τον πρώτο, είναι ότι ο συγκεκριμένος κλάδος θα πρέπει να γίνει πιο ανθεκτικός, ικανότερος δηλαδή να ανθίσταται στα σοκ. Και ταυτόχρονα ε, ο ίδιος ο τομέας αυτός να διατρέχει λιγότερους κινδύνους. Ξέρουμε όλα αυτά τα οποία λένε τράπεζες όπως η BNP, η Paribas, η Barclays κτλ. Λένε ότι θέλουν να έχουν για τους μετόχους τους 20% απόδοση. Για ακούστε λίγο. Σε μια λειτουργούσα έβριθμα την αγορά τέτοιου είδους κέρδη δεν είναι δυνατό να υπάρξουν διψήφια εκτός αν υπάρξει στρέβλωση της αγοράς, ασυμμετρία ενημέρωσης και έλλειψη διακανονισμών. Δεν είναι λοιπόν αυτό το σημάδι σημάδι καλό αυτά τα κέρδη αυτά λοιπόν δεν είναι εφικτά. Και δεν το λέω αυτό γιατί ιδεολογικά εμείς θα θέλαμε να υπάρξει μια διαφορετικού τύπου λειτουργούσα αγορά. Αλλά τα κεφάλαια τα οποία πηγαίνουν στη χρηματοπιστωτική αυτή ε, δραστηριότητα δεν πηγαίνουν στην πραγματική παραγωγή, στην πραγματική βιομηχανία, στο πραγματικό λιανεμπόριο, το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα έβρεσης χρηματοδότησης και κεφαλαιοποίησης. Αυτό από, από πλευράς του χρηματοπιστωτικού τομέα συνιστά θα έλεγα στρέβλωση του ανταγωνισμού. Απαιτείται λοιπόν ισορροπία με τον τομέα, με τον κλάδο αυτό. Το να προσπαθήσει κανείς με μία νομική ρύθμιση να υπερασπιστεί όλα τα νομικά πρότυπα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτείται να υπάρχει μία ποικιλία θα έλεγα στα business models τα οποία επιδιώκουμε. Καταλαβαίνω βέβαια αυτά τα οποία είπατε πρόεδρε να βασιστούμε κατά βάση στην ε, έκθεση πρωτοβουλία που ψηφίσαμε πέρυσι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Και ίσως αυτά τα οποία πιστεύαμε πριν έξι μήνες ότι δηλαδή ε, τα μέτρα που θα λαμβάναμε τότε είναι επαρκή, τώρα δεν ισχύει. Και θα ήθελα να προκαταλάβω ίσως και κάποιες αντιρρήσεις τις οποίες ακούμε από πλευρές. Μην είστε σκληροί προς την οικονομία μας λένε. Στην παρούσα φάση η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και με τους κανόνες και χωρίς τους κανόνες της Βασιλείας 3 δεν υπάρχει ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις. Εκτός από κάποιες νης, κάποιες, ε, κάποιους πολύ μικρούς τομείς που θεωρούνται ασφαλείς όπως η ενέργεια γιατί οι τράπεζες λένε «Α, αυτό είναι επικίνδυνο» ή «Το άλλο είναι επικίνδυνο». Ας μην επιλέγουμε λοιπόν ε, το επιχείρημα ότι αν είμαστε αυστηροί δεν θα μας δανείσουν. Όχι, είναι πιο απλό. Δεν μας δανείζουν, τίποτα άλλο. Δεύτερον, δεύτερο επιχείρημα το οποίο ακόμη μην είστε πολύ σκληροί γιατί στην ουσία θα καταστήσετε ασθενέστερη την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαϊκών Πιστοτικών Ιδρυμάτων. Όταν βλέπω την κατάσταση βλέπω ότι πολλέ από, ε, από τα Ευρωπαϊκά Πιστοτικά Ιδρύματα είναι εξασθενημένα, χωρίς περαιτέρω κανόνες. Και πιστεύω ότι οι σκληροί και οι ε, <clears throat> σωστοί κανόνες θα τις θα τα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικά. Και σχέση τώρα με το level play field, δηλαδή το να ξεκινήσουν όλοι από το ίδιο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είναι προς το καλύτερο συμφέρον της ευρωπαϊκής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις τις οποίες θα ήθελα να κάνω για να περάσω ίσως σε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με το επίπεδο των κεφαλαίων, κεφαλοχή επάρκεια. Νομίζω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία εγώ έχω, είμαι μηχανικός που έχω ειδικευτεί σε μαθηματικά μοντέλα. Ξέρω τις αδυναμίες αυτής της δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν αυτό το benchmark το οποίο θες να χρησιμοποιείτε για την αντιμετώπιση και αξιολόγηση του επίπεδου κινδύνων είναι χρήσιμο. Από την άλλη δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι μπορούμε να εξαρτηθούμε απόλυτα από τέτοιου είδους μοντέλα διαχείρισης κινδύνου και να μην ζητήσουμε τα επίπεδα, τα κεφαλογικά να είναι υψηλότερα από αυτά τα οποία απαιτεί η Βασιλεία 3. Εγώ εδώ συμφωνώ περισσότερο με το Λονδίνο από ότι με την υπόλοιπη Ευρώπη ίσως. Μη μου λέτε ότι τα υψηλότερα κεφάλαια σώζουν την οικονομία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό θέλω να διαπραγματευθώ με τις α, τράπεζες αλλά όχι με αυτές ιδιαίτερα τις μεγάλες οι οποίες λένε ότι αυτό το επιχείρημα είναι αυτό το οποίο τις οδηγεί στο να μην δανείζουν χρήματα. Αυτά είναι ανοησίες. Ταυτόχρονα σε σχέση με το, με το μοντέλο κινδύνου, αξιολόγησης κινδύνου αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η μη έκθεση στον κίνδυνο και Νομίζω ότι το κείμενο λέει πάρα πολλά θετικά, ιδιαίτερα σχετικά με τη μόχλευση. Uh, liquidity is... well, we have... Ναι, και ισχύει φυσικά και για την περίπτωση της ε, Γαλλοβελγικής Τράπεζας Δέξια. Πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες σε σχέση με τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ε, όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν πριν μερικές εβδομάδες για τις γελικές τράπεζες είχαν σχέση με τη ρευστότητά τους. Έχουμε την πολυτέλεια λοιπόν να περιμένουμε 3, 5, 4 χρόνια για να επιβάλλουμε κάποια επίπεδα υποχρεωτικής ρευστότητας. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει σήμερα. Η έλλειψη ρευστότητας είναι κάτι το οποίο απειλεί σήμερα. Ας μην πειραματιζόμαστε λοιπόν. Καιρό είναι λοιπόν να πάρουμε μέτρα τώρα, τώρα για τα business models. Όσο κοιτάω αυτές τις προτάσεις, Και εδώ η έκθεση της Βίκη ήταν καλή. Έχει σημασία να έχουμε υδατοστεγή, αν θέλετε, ε, διαμερίσματα τα οποία να μπορούν να αντέξουν τα οικονομικά σοκ και να διασφαλίσουμε την δυνατότητα των μεγάλων πιστοτικών ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο των ευρωπαϊκών. Να μην βλάπτουμε, γιατί αυτό κάνουμε σήμερα, την ικανότητα της οικονομίας μας να ταξιδέψει στους ωκεανούς. Κάποιες λεπτομέρειες που νομίζω ότι έχουν κάποια σημασία. Όταν θα συζητάμε εμείς το CRD4, οι κανόνες για τα θεσμικά ιδρύματα τα οποία είναι πολύ μεγάλου μεγέθους για να πτωχεύσουν ή να αποτύχουν θα έχουν ήδη κυκλοφορήσει πριν το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα τη χρονική να συμπεριλάβουμε ε, τα ειδικά χαρακτηριστικά για τα πολύ μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα σε αυτές τις προτάσεις. Κοιτάξτε, κάνουμε ένα αγώνα με το χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό το too big to fail, πολύ μεγάλο για να αποτύχει, είναι θέμα υπαρξιακό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποια πιστοτικά ιδρύματα να μας εκβιάζουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στο CRD4. Και τέλος το τελευταίο θέμα είναι η μεταβατική περίοδο. Ακόμα και όταν είναι κανείς ιδιαίτερα στραμμένο στα μακροπρόθεσμα, το 2019 είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2019 για τον εξασθενημένο ε, χρηματοπιστωτικό τομέα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηρότεροι κατά τη διάρκεια αυτή τη μεταβατική περίοδου. Πρέπει να είναι συντομότερη αυτή η μεταβατική περίοδο και να έχουμε συγκεκριμένα κίνητρα έτσι ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω αναμονή. Να αυξηθεί η διαφάνεια και σε σχέση με τον έλεγχο τη ρευστότητα, να είναι δημόσια διαθέσιμε οι πληροφορίε για τη ρευστότητα των πιστοτικών ιδρυμάτων και σήμερα όμω τώρα και όχι να περιμένουμε στο μέλλον για να γίνει κάτι τέτοιο γιατί θα πρέπει να έχουν την επιλογή είτε να κλείσουν την πόρτα τους είτε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους τα πιστοτικά ιδρύματα. Είναι ένας αγώνας λοιπόν εναντίον του χρόνου. Δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία για να προφλάσουμε ε, τις καταστροφές που ε, θα έλθουν αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους σκιώδεις εκτός ο Γκούναρ έχει το λόγο τώρα. Από το ΕΛΚ δεν είναι παρόν Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε ο για το παράδοξο αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες μπορούν να δανείζουν περισσότερο. Αλλά συγχρόνως στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι μαζεύονται στο καβούκι τους και δανείζουν λιγότερο. Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν αυτή την νομοθεσία είναι απαραίτητο να τη θέσουμε την νομοθεσία αυτή σε ένα γενικότερο πλαίσιο θεμάτων που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. είναι απαραίτητο καταρχήν να μην ξεχάσουμε τη σημασία της στάθμισης κινδύνου. Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της μόχλευσης ο Φίλιπ, <clears throat> αλλά σε τελική ανάλυση το απαραίτητο είναι να κρατήσουμε την ιδέα της στάθμισης κινδύνων, γιατί αν δούμε τις διάφορες χρηματοπιστωτικέ αγορές, είναι πραγματικά μεγάλε οι διαφορέ οι οποίε υπάρχουν. Βλέπετε παραδείγματο χάρη την κατασκευαστική βιομηχανία από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά τι νέε επιχειρήσει στο βιομηχανικό τομέα και στι υπηρεσίε. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην ξεχάσουμε την πολυμορφία που υπάρχει στα, στις δραστηριότητες αυτές και να έχουμε μια σωστή στάθμιση κινδύνων. Το επόμενο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι κάτι το οποίο πιστεύω πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε στη συζήτηση, συγκεκριμένα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι τράπεζες πρέπει να δείξουν από μόνες τους την ε, πρέπουσα φροντίδα και την ε, ε, υπευθυνότητα. Ακόμα και δεν είχαμε κεφαλαιοχικές απαιτήσει καθόλου σε ρυθμιστικό επίπεδο. Είναι προφανώς προς το συμφέρον των τραπεζών να αναλάβουν μόνες τους την ευθύνη να έχουν κάποια αποθεματικά. Ξέρουμε βέβαια όλοι ότι οι τράπεζες θεωρούν ότι θα είναι αιώνιες θα δουλεύουν στο Δινεκές, γιατί αν πάει κάτι στραβά θα έρθουν τα κράτη και οι κυβερνήσει και θα τις διασώσουν. <clears throat> Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν συζητάμε για τα θέματα επίλυσης τραπεζικών προβλημάτων. Αλλά μέσα στα πλαίσια αυτή τη νομοθεσία πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζε από μόνε του θα φέρονται με ένα υπεύθυνο τρόπο. Η τρίτη μου παρατήρηση είναι η εξή. Έχουμε μόλι εγκρίνει το νέο σύμφωνο σταθερότητος. Είναι και εδώ πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορούμε να θέσουμε ότι επίπεδο κεφαλουχικών απαιτήσεων θέλουμε, αλλά χωρίς μακροοικονομική σταθερότητα όλα αυτά είναι άχρηστα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό το πλαίσιο μακροοικονομική σταθερότητα και ότι θα έχει κάποιο αντίκτυπο. Το λέω αυτό γιατί πολλέ φορέ μιλάμε για κεφαλουχικέ απαιτήσει και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα αυτοσκοπό, ότι αυτό είναι κάτι απομονωμένο από όλα τα άλλα <clears throat> ζητήματα. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματικότητα. Για την έκθεση αυτή που έχουμε ενώπιον μας σήμερα νομίζω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και ένα άλλο τμήμα της πραγματικότητας ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα από ό,τι σε άλλες. Και ο δανειστής, το να είναι κανείς δανειστή τελευταία καταφυγή, αυτό δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη στις κυβερνήσει των χωρών αυτών από ότι στις χώρες που η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα είναι πιο μικρή σε έκταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι όταν αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε ορισμένε χώρε, εάν το επιθυμούν, να έχουν υψηλότερε κεφαλουχικέ απαιτήσει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια, όπου τα κράτη-μέλη ή γενικά τα κράτη της Ευρώπης είχαν ιδιαίτερα ε, διογκωμένους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Το πιο εξόφθαλμο παράδειγμα είναι ίσως η Ισλανδία. Και φυσικά η νομοθεσία περί των τραπεζικών θεμάτων στην Ισλανδία θα μπορούσε να είναι διαφορετική από ότι η τραπεζική νομοθεσία στην ε, Γαλλία σε ό,τι αφορά το επίπεδο κεφαλαιογικών ε, απαιτήσεων λόγω του μεγέθους του τομέα αυτού. Θα πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Όσο λοιπόν δεν αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα να επιβάλλει κάποιο υψηλότερε απαιτήσει κεφαλογικού χαρακτήρα στα κράτη-μέλη όπου ο χρηματοπιστωτικό τομέα έχει ιδιαίτερη εμβέλεια. Ευχαριστώ. Ο Διέγκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σάρων. Θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντα τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, την Αλή Μακάρθη, τον τρόπο με τον οποίο επίσης εργάστηκε στην έκθεση πρωτοβουλία της και φυσικά θέλω να ευχηθώ καλή τύχη για την πολύ δύσκολη εργασία που έχουμε ενώπιόν μας τους επόμενους μήνες. Κάποιες παρατηρήσεις για τα θέματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Με την εισαγωγή του συστήματος της Βασιλείας 3, οι κανόνες για τις κεφαλογικέ απαιτήσει και τη ρευστότητα των τραπεζών υφίστανται σημαντικές τροποποίησεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητες αυτές οι τροποποίησεις και αυτό αναφέρθηκε ήδη, αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να συνδέσουμε αυτές τις αλλαγές με την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας και να καταλάβουμε ποιες είναι οι συνέπειες και οι απόρριες αυτών των νέων μέτρων στον τραπεζικό τομέα στην πραγματική οικονομία των κρατών μελών. Υπάρχουν ορισμένα αριθμητικά στοιχεία τα οποία εγώ είδα για την πορτογαλική οικονομία και ίσως αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε κι εσείς. Η εφαρμογή απλώς και μόνο των κανόνων της Βασιλείας θα οδηγήσει σε αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική ανάπτυξη της Πορτογαλίας σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ σε μακροχρόνιο επίπεδο. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει και σε μια όξυνση της ανεργίας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Απόλυα 7 με 7.5 χιλιάδων θέσεων απασχόλησης και σε ό,τι αφορά την πιστοτική αγορά προβλέπεται μια αύξηση κατά 3% σε μακροχρόνιο επίπεδο όταν η αρχική πρόβλεψη χωρίς τους κανόνες Βασιλείας 3 ήταν 6,2. Και επίσης προβλέπεται για τα, την επιβάρυνση επιτόκια από 0,9 να φτάσουν το 3,1%. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προβληματική αυτή θα πρέπει να γενικεύσουμε την προβληματική, να δούμε τι θα γίνει στα διάφορα κράτη-μέλη με την εισαγωγή της Βασιλείας 3 και επίσης θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε το ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πλήρως τους κανόνες της Βασιλείας 3 και θα προσεγγίσουν με τον τρόπο αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο. Γιατί ξέρετε ότι η μη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έθιξε σημαντικά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και έμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία. Για να κλείσω. Η τρίτη μου παρατήρηση είναι η εξή. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν ορισμένε περιοχέ οι οποίε έχουν ιδιαίτερη, ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα και σε σχέση με του οποίου εγώ έχω παρουσιάσει κάποιε τροπολογίε στην έκθεση πρωτοβουλία και θα το πράξω και στην τρέχουσα νομοθετική έκθεση. Υπάρχουν προβλήματα στο πορτογαλικό νομικό σύστημα. <clears throat> Αναφέρομαι στα συνταξιδοτικά ταμεία, στην διαφύλαξη των συμφερόντων των μειοψηφίων, μη μειοψηφιών, στο αποθεματικό κεφάλαιο με σε εισαγωγικά μαξιλάρι, που προστατεύει την κεφαλογική βάση, και επίσης την ανάγκη να διατηρήσουμε την πρόσβαση, την απρόσκοπτη πρόσβαση στα στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα παραγνωρίσουμε, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μας ιδιαίτερα όταν θέλουμε να δούμε τη σύνδεση μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και, του, και της πραγματικής οικονομίας που έχει τόσο μεγάλη σημασία για την Ευρώπη. <coughs> Ευχαριστώ, λέει. Η, ο, όλοι έχει το λόγο. Η Αρλίν μάλλον. Ναι, σύμφωνα και εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη υποστήριξη στον εισηγητή μας στα θέματα αυτά. Είναι πεπλεγμένα θέματα, αλλά είναι και πολύ δύσκολη η καιρή και είναι πολύ δύσκολο να βρει κανεί την σωστή ισορροπία. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο σε ορισμένε γενικέ ε, ε, και θα αφήσω του εμπειρογνώμονε που έχουμε πολλούς στην Επιτροπή μα. Είναι πολύ καλό ότι έχουμε εμπειρογνώμονε σε αυτά τα θέματα να αντιμετωπίσουν τα πιο λεπτομεριακά θέματα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μειώσουμε <clears throat> την, ε, ε, τον κίνδυνο κρίσεων και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τι κρίσει. Πιστεύω ότι μπορούν να πτωχεύσουν οι τράπεζε, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε καταράκωση τη οικονομία και σε ζημιά στου ε, πολιτέ και του καταναλωτέ. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρε εμένα ω εισηγήτρια για τι κεφαλαιοχικέ απαιτήσει 3, CRD3, είναι ότι κινδυνεύουμε να δούμε τις τράπεζες να ζητάνε να υπάρχουν πιο ασθενείς κανόνες, να υπάρχουν αναδιατάξεις και επανυπολογισμοί, όπως είπαν και πολλοί από τους ε, <clears throat> εμπειρογνώμονές μας, Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα και να υπάρξουν ανεξάρτητες μελέτες και επαληθεύσεις. Γιατί αυτό το οποίο περιέχουν οι προτάσεις CRD4 είναι ένα σχέδιο 10 ετών. Μέσα σε 10 χρόνια μπορεί κανείς να εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων. Τέσσερα χρόνια μετά την έκρηξη της κρίσης η τράπεζές μας είναι ακόμα σε πολύ δύσκολη θέση και οι οικονομίες μας πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Δεν <clears throat> φτάνουν όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει από μόνα τους και να ξεπεράσουν την κρίση. Βλέπετε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Η έκθεση της Τράπεζας της Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι στο 4ο τέταρτο του 2011 ε, υπήρξε μια αύξηση των διαθεσίμων των τραπεζών κατά 5 δισεκατομμύρια ε, λίρε, αλλά παρόλα αυτά δεν αυξήθηκε ο δανεισμό. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν αυτό, εφόσον έχουν λεφτά οι τράπεζε γιατί δεν τα δανείζουν. Είδατε πολύ αυτά που είπε ο Τζορτ Όσουελ, ο, ο επικεφαλής της τράπεζας της Αγγλίας χθε, είπε ότι και πάλι θα ρίξει το μπαλάκι στον φορολογούμενο και θα αφήσει τι τράπεζε χωρίς να παίρνουν κανένα κίνδυνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας να δούμε αν οι τράπεζε πράγματι δανείζουν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Να έχουμε μια μελέτη για τα θέματα αυτά. Σάρων πρέπει να επιστρέψουμε και να εξετάσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου, δεν έχουμε ιδέα αν οι τράπεζε πράγματι δανείζουν στι μικρομεσαίε και ποια είναι η κατάσταση. Επομένω, εγώ <clears throat> υποστηρίζω, εκτό αν υπάρχει αποχρόν λόγο, να εφαρμόσουμε πλήρω τη Βασιλεία. Η μελέτη που κάναμε τον Ιούλιο, που ζητήσαμε να γίνει τον Ιούλιο, δείχνει ότι μπορεί κανείς να αυξήσει τις κεφαλογικές απαιτήσει μέχρι τα 13% κιόλα, περισσότερο από ό,τι λέει η οδηγία, χωρίς κάποιο κίνδυνο για την πραγματική οικονομία ούτε για τις τράπεζες. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω, που είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει αυτά που είπε ο κύριος Χέρκμαρκ. Εγώ ανησυχώ για την προσέγγιση βάση εναρμόνισης. γιατί δεν θέλουμε να έχουμε υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις κεφαλογικές απαιτήσει. Ένα αγώνα προς τα άνω, όχι προς τα κάτω. Λένε ορισμένοι ότι αυτό θα οδηγήσει σε στρέβλωση τη εσωτερική αγορά. Αλλά συγχρόνω, όλοι μα θέλουμε να έχουμε υψηλότερε κεφαλογικέ απαιτήσει, ασφαλέστερη αγορά, να μπορούν οι τράπεζε πραγματικά να δανείζουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό όμω δεν σημαίνει να, προ... να κατέβουμε σε ό,τι αφορά τα πρότυπά μα, να μειώσουμε τα πρότυπά μα το θέμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο δικό μου κράτος μέλος είναι ότι έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση η οποία όμως δεν οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαιοχικών απαιτήσεων για τις τράπεζες που δανείζουν στον καταναλωτή ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στην περίπτωση αυτή που θα υπάρξει μια κρίση θα προστατευτούν οι καταθέσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες δανείζουν. Γιατί δεν αυτό λοιπόν στρέβλωση στην ε, ενιαία αγορά. Γιατί με το σύστημα του διαβατηρίου μέσα εισαγωγικά ξένες τράπεζες μπορούν να λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να υπόκεινται στους αυστηρούς περιορισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου για τα, τις κεφαλογικές απαιτήσει για την μικρή κλίμακος τραπεζική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε υψηλά στάνταρ και υψηλέ κεφαλογικέ απαιτήσει, ότι δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Αυτό δεν αποδεκτό. Νομίζω πρέπει να έχουμε μια πιο εφάνταστη αντιμετώπιση στην ε, Επιτροπή μα. Αυξάνεται ο κατάλογο των αγορητών, αλλά υπάρχει και πρόβλημα χρόνου για τη σημερινή συζήτηση. Επομένως, εάν χρειαστεί θα σας ε, περικόψω. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος, να το Ο έχει Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Äh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον Ότμαρ Κάρας για την εξαιρετική εργασία του. Ακριβώς η οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις, η τέταρτη γενικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ τεχνική όσο και σημαντική. Ε, σήμερα το πρωί να κάνω μερικά σύντομα σχόλια. Καταρχήν, καλωσορίζω τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποσοτικά και ποιοτικά. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι μεγαλύτερε οι κεφαλαίκε απαιτήσει. Το είδαμε τους τελευταίους μήνες άλλωστε και το ζήσαμε και μα το έδειξε και η κρίση. Σίγουρα θα υπάρξει ε, και κάποια αντίδραση των τραπεζών στην προσαρμογή στην νέα κατάσταση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αντανακλάται στις χορηγήσεις. Το είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ρητά εδώ και τη δανειοδότηση του δημοσίου. Γι' αυτό και αυτή είναι μεγάλη αποστολή και το καθήκον της ε, Επιτροπής μας, ε, θα πρέπει τους κανούς αυτούς να τους διατυπώσουμε όσο γίνεται πιο προσεκτικά. Καλώς ορίζω τον ουδέτερο ορισμό ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το βασικό κεφάλαιο και τις ρυθμίσεις για την προστασία και τις μεταβατικές. Δεν ξέρω κατά πόσο αρκούν, θα το ελέγξουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τις μικρότερα σε ποσοστά ε, μερίδες συμμετοχή Θα το κοιτάξουμε και το ίδιο για τη ρευστότητα, αλλά και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της EBA, στο σύστημά μας. Πολλές ρυθμίσεις που παραπέμπουμε σε αυτή την αρχή δεν είναι μόνο τεχνικές, αλλά κατά την άποψή μου έχουν και πολιτική υφή και θα πρέπει κατά τη διάρκεια των επόμενων συζητήσεων να τα κοιτάξουμε αυτά και σε λεπτομέρειες. Ε, και ε, το τελευταίο είναι ε, οι λόγοι κατανομής σε διάφορα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει σχεδιάσει, αλλά αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες δυσκολίες σχεδιασμού και προγραμματισμού τη επιχειρήση. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, πολύ τηλεγραφικά σημεία. Τις επόμενες εβδομάδες σίγουρα θα έχουμε να κάνουμε αρκετά, αλλά είμαι βέβαιος, ότι θα τα καταφέρεις και εσύ και τα μέλη της Επιτροπής θα βοηθήσουν ε, και θα συνδράμουν όπως αρμόζει τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια γενική παρατήρηση και μια κάπως πιο συγκεκριμένη. Ακούγοντας το Φιλίπ, ο οποίος δυστυχώς έφυγε, έχει ένα εξαίρετο τρόπο να παρουσιάζει τις απόψεις του ο Φίλιπ. Το είχα πει και πριν. Εμείς χρειαζόμαστε τράπεζες που να έχουν καλή υγεία στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχει κανείς αποτελεσματικές και λειτουργικές ε, υγιείς τράπεζες στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να κυνηγάμε και να κατηγορούμε και να χτυπάμε τις τράπεζες σαν να ήταν η μοναδική μας δραστηριότητα εδώ. Μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική στις τράπεζες και σωστά ίσως, αλλά πολλά από τα λάθη αυτά έχουν γίνει από τους πολιτικούς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες και κάποιοι από αυτούς, μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε και πρόεδρος. Δεν τα έλεγε αυτά πριν γίνει πρόεδρος. Και πολλοί από τους γερουσιαστές το ίδιο και αυτοί δεν έλεγαν πραγματικά τι συμβαίνει γύρω από όλα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να σκεφτούμε την κατάσταση απέναντι στις τράπεζες και να είμαστε, ε, να κάνουμε και αυτοκριτική, όχι μόνο να κατηγορούμε τις τράπεζες. Η βασική μου παρατήρηση τώρα. Συμφωνώ με τον Γκούναρ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνει όλες τις χώρες να έχουν τους ίδιους κανονισμούς και τους ίδιους κανόνες. Αν μια χώρα θέλει αυστηρότερους κανόνες, δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι τέτοιο επηρεάζει αρνητικά τις άλλες χώρες. Είναι ένα σύνδρομο αυτομαστίγωσης αν θέλετε αυτό. Δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση το ότι δεν σεβόμαστε τους κανόνες του ανταγωνισμού και αν υπάρχουν κάποιες αρνητικές εμπειρίες σε ορισμένες χώρες και αυτό έχει υπάρξει τα τελευταία 20-25 χρόνια θα πρέπει να το σκεφτούμε και να είμαστε πιο σε εισαγωγικά φιλελεύθεροι και να επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να έχουν ισχυρότερους και αυστηρότερους κανόνες αν ο τραπεζικός τομέας στις χώρες αυτές είναι πολύ μεγαλύτερος και σημαντικότερος σε σχέση με το ΑΕΠ Ελπίζω να υπάρξουν κάποιες τροπολογίες και ελπίζω και εσείς να σκεφτείτε ότι το επιχείρημα αυτό έχει νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σβέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ μια ακόμα φορά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Όθμαρ Κάρας για την τεράστια εργασία που έχει επενδύσει και σε αυτή και στην προηγούμενη έκθεση. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν που μας έχει δώσει την απαραίτητη τεκμηρίωση. Για πάρα πολλούς από τους πολίτες μας, το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί η κρίση διαρκεί τόσο πολύ καιρό. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έκδηλο. Τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, σε ό,τι αφορά τους ε, κοινούς κανόνες, Μπορεί να έχουμε δεχθεί τη Βασιλεία Τρία, αλλά η πραγματική εφαρμογή των κανόνων και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα αντιμετωπίζει μεγάλα προσκόμματα. <clears throat> και αυτή τη στιγμή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ επισφαλής. Έχουμε λοιπόν ένα διπλό πρόβλημα. Καταρχήν είναι ένα πολύ, πολύ πλοκό πλέγμα κανόνων και συστημάτων που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς και από την άλλη πλευρά υπήρξε μια καθυστέρηση στην εφαρμογή όλων αυτών των ε, κανόνων. Εγώ χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δεν έχει καθυστερήσει, αλλά έθεσε τις απαιτήσει της για πιο αυστηρά πρότυπα, τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε διεθνές επίπεδο ακόμα. Το πραγματικό ερώτημα, το οποίο όμως εγώ θέλω να θέσω από τη δική μου πλευρά, είναι πέραν της γενικής συνένεσης ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα ίδια κεφάλαια στις τράπεζες, να υπάρχουν περισσότερο, πόσο και για ποιου θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κεφάλαια. Από τη δική μα πλευρά, το ίδιο κεφάλαιο των πιστοτικών ιδρυμάτων εξακολουθεί, οι απαιτήσει οι οποίε ισχύουν ακόμα και τώρα, εξακολουθούν να είναι χαμηλέ, πολύ χαμηλέ. Αν αντιμετωπίσουμε λοιπόν σωστά το θέμα, θα πρέπει να το συνδέσουμε και με την χρηματοδότηση, με τις χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία οι τράπεζες οι οποίες δανείζουν στην πραγματική οικονομία έχουν πραγματικά μια, υγεία, μια υγιή οικονομική κατάσταση. Αντίθετα από αυτές που έχουν ε, πολύ μεγάλη μόχλευση και δεν κάνουν τίποτα τέτοιο. Όπως είπε ο Μάρτιν Χέλβικ, ο επικεφαλής του, συστημικού, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και οι αρμόδιοι της ε, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη κεφαλαιογική απέτηση. Και βλέπει κανείς ότι χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ελβετία που έχουν φυγεί ιδιαίτερα από την κρίση ζητούν τώρα να υπάρχουν μεγαλύτερες κεφαλαιοχικές απαιτήσει. Κατά δική μου άποψη λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε και ένα δεύτερο ερώτημα. Να έχουμε μια πραγματικά σκεπτικιστική αντιμετώπιση σε σχέση με την εκτίμηση του κινδύνου μέσω εσωτερικών ε, μοντέλων όπως επιτρέπει η Βασιλεία πόσες είναι οι τράπεζες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα με εσωτερικά μοντέλα να κάνουν σωστή αξιολόγηση κινδύνου και πόσες τράπεζες έχουν διοικητικά συμβούλια τα οποία είναι σε θέση να ελέγξουν ότι πραγματικά γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα αποθεματικά που έχουν οι, οι τράπεζες είναι το τελευταίο προπύργιο πρώτης ε, κατάρρευσης. Όταν δεν έχουμε όρια μόχλευση όπω ίσχυαν στο παρελθόν στι ΗΠΑ, αυτό είναι το τελευταίο όριο. Είδαμε λοιπόν στην κρίση ότι πάρα πολλοί κίνδυνοι στην αρχή δεν φαίνονται καν ότι είναι κίνδυνοι. <clears throat> Ένα από τα αγαπημένα θέματα αυτά είναι το, η μηδενική στάθμιση κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα. Πριν από μερικά χρόνια αυτός το θεωρού, ο κόσμος το θεωρούσε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Αυτός είναι όμως και ένας από τους μεγάλους ε, ε, λόγους για τους οποίους πρέπει να έχουμε επιπροσθέτως και ένα ανώτατο όριο μόχλευσης, γιατί δεν μπορούμε πάντα τους κινδύνους αυτούς που δεν τους διαβλέπουμε να τους αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε αρκετά ίδια κεφάλαια. <clears throat> Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια πιο ισχυρή βάση κεφαλαιακής ε, επάρκειας, θα πρέπει να δούμε και τη σχέση αυτών των κεφαλαίων με την χορήγηση στην πραγματική αγορά. Και επομένως θα πρέπει να κάνουμε διάκριση διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων για διάφορες μορφές τραπεζικών δραστηριοτήτων και να μην έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία ενιαία για όλους. Έχουμε λοιπόν το, την οδηγία για την κεφαλογική επάρκεια 2 και 3, αλλά δεν έχουμε ακόμα <clears throat> την ε, οδηγία για τα συστημικά <clears throat> θέματα κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες να, όταν έχουμε κανόνες οι οποίοι αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγχρόνως τις μεγάλες επιχειρήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει και οι, οι που έχουν μεγάλη σημασία για την, ε, σε ό,τι αφορά την ε, συλλογή φορολογικών εσόδων και αυτές να λαμβάνονται υπόψη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια των κανόνων και να βρούμε τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μεταβιβάζεται, δεν μετακυλίζεται η ευθύνη πάντα στα κράτη. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αντιμετωπίσω είναι το θέμα της λεγόμενης σκιώδους τραπεζικής δραστηριότητας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ρυθμίζουμε τις υπηρεσίες, τις τράπεζες οι οποίες χορηγούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αφήνουμε τελείως αχαλήνοτη την δραστηριότητα ε, τραπεζικών φορέων σε άλλες δραστηριότητες. Δυστυχώς το είδαμε αυτό και στη συζήτηση για τα hedge funds, για τα ταμεία αντιστάθμισης. Δεν μπορέσαμε να έχουμε μια συμφωνία για τις ε, υποχρεώσεις τους σε ίδιο κεφάλαιο Πρέπει να έχουμε όμως κάποια ρύθμιση στον τομέα του shadow banking, της σκιώδους τραπεζικής δραστηριότητας, αλλιώς θα έχουμε μία, μία ανισότητα ανταγωνισμού. Δεν μπορούν οι τράπεζες να υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση και όχι τα hedge funds. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο επίσης είναι το θέμα της αναλογικότητας. Θα μπορούσε για τους ίδιους κανόνες, αν τους εφαρμόσουμε με τον ίδιο τρόπο, σε τράπεζες οι οποίες έχουν την παραδοσιακή, τη λεγόμενη βαρετή διαδικασία τραπεζικής, μπορούν μικρές ε, τράπεζες να πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο χαρτοβασίλειο υποχρέωσεων <clears throat> παραγωγής αναφορών κτλ. που ισχύει και για τις μεγάλες τράπεζες. Ο Ότμαρ Κάρες νομίζω το έχει θίξει αυτό το θέμα, ότι πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη αντιμετώπιση και επίσης ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο νόμος θα έχει ένα ουδέτερο χαρακτήρα και δεν θα πλήττει περισσότερο ορισμένες μικρότερες τράπεζες. Εμένα με ενοχλεί πάντως η ιδέα να φέρουμε σε εφαρμογή αμέσως αυτούς τους κανόνες που αυτό απαιτεί την εκπόνηση τουλάχιστον 150 παραγόγων αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Αν λοιπόν σπρώχνουμε όλα αυτά τα νομοθετήματα και τις ρυθμίσεις με τέτοια ταχύτητα, τότε οι μικρές τράπεζες που δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό δεν θα είναι σε θέση να μπορέσουν να εφαρμόσουν όλη αυτή την νομοθεσία και τις ρυθμίσεις και το αποτέλεσμα θα είναι τελικά ότι το λόμπι των μεγάλων ε, τραπεζών θα τρίβει τα χέρια του γιατί θα έχει βγάλει τις μικρές ε, τράπεζες από το παιχνίδι. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να τονίσουμε ότι χρειάζεται περισσότερο ε, ίδιο κεφάλαιο, δεν πρέπει να το αφήνουμε να το εκτιμούν μόνο οι τράπεζες με τα δικά τους μοντέλα, αλλά επίση πρέπει να έχουμε και κάποια μέτρα τα οποία θα είναι διαφοροποιημένα, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς οι οποίες ε, κινδυνεύουν από την υπερβολική ρύθμιση και την υπερβολική νομοθεσία και συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι τα, τα θύματα κρίσεων. Ορισμένοι λένε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι προϊόντα αρπαγής, ότι υπάρχει μια αρπακτική στάση των τραπεζών στα θέματα αυτά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία δεν εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση της αγοράς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πραγματικά με, τον, με τη σωστή θέση του νομοθέτη και όχι να αφήσουμε τις τράπεζες να αλωνίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι εμπιστεύομαι τον εισηγητή τον κύριο Κάρας και τις ικανότητές του να βρει μια ισόρροπη λύση. Τρία είναι τα θέματα που με ανησυχούν. Πρώτον, η ανάγκη να υπάρξει μια συνολική συνοχή στον τρόπο με ε, τον οποίο χειριζόμαστε τις κεφαλικές απαιτήσει. Δεύτερον, η ανάκαμψη της οικονομίας και τρίτον, είναι ευρωπαϊκή λύση. Πρώτον, η συνολική έτσι, συνέπεια και συνοχή. Αξίζει να αναφερθούν τα εξή στοιχεία. Η Ευρώπη είναι ηγέτης παγκοσμίω στο τραπεζικό σύστημα. 75% της μεσολάβησης ε, γίνεται ε, στις τράπεζες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ε, στις χρηματαγορές. Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό, να παραμείνει η δραστηριότητα αυτή τραπεζική και να μην περάσει στα χρηματιστήρια. Ε, δεύτερον, ο τομέας εφαρμογής. Μόλις γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βασιλεία 3 αφορά 20 τράπεζες, ενώ στην Ευρώπη 8.000 ε, ιδρύματα. Στην Ευρώπη θέλουμε κάτι που να ισχύει για όλα τα πιστοτικά ιδρύματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάποια αναλογικότητα όντως και κάποια λογική για να μην παίζουμε από μια νοικτική θέση. Επόμενο θέμα, να είναι ουδέτερο το σύστημα και το μοντέλο ε, ε, συναλλαγών θα πρέπει να είναι νέο ε, στην Ευρώπη να μην τιμωρούνται οι μικρομέτωχοι γιατί οι ίδιοι ε, βάζουμε εμπόδια στον εαυτό μας και θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά τα θέματα. Συνοχή, ε, ο τομέας εφαρμογής και ουδετερότητα. Δεύτερον, οικονομία και ανάκαμψή της. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται βαθιά μεταρρύθμιση στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτή για να είναι συμβατή με την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση ίσως θα πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο τις απαιτήσει μας και είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητηθεί και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Και ένα τρίτο στοιχείο, η ευρωπαϊκή διάσταση. Γίνεται λόγος για πλήρη εναρμόνιση. Εγώ είμαι πάντα υπέρμαχος ευρωπαϊκών προτύπων που να δείχνουν ένα επίπεδο εμπιστοσύνη σε όλη την Ευρώπη για όλες τις δραστηριότητε, αλλά πιστεύω επίσης ότι πρέπει να υπάρχει και κάποια δυνατότητα. Δεν λέω τα κράτη-μέλη να βάζουν διαφορετικές απαιτήσει, αλλά ανάλογα με τον κίνδυνο κάθε κράτος μέλος να ορίζει κάποιες απαιτήσει, ενδεχομένως υψηλότερε, αλλά που να εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο εντό του κράτους, αλλά όπου υπάρχει κίνδυνο. Δηλαδή όλα τα ιδρύματα που λειτουργούν σε ένα κράτος και όλες οι υποπτικές αρχές. Και αν κάποιος θεωρεί ότι είναι δυσανάλογα, ευτυχώς σήμερα έχουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και ένα σύστημα εποπτείας για να λύνει τέτοιου είδους προβλήματα. Ευχαριστώ. Η Ελίσσα. Ευχαριστώ, Σάρων. Και εγώ θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στον Ότμαρ Κάρας για το έργο που έχει φέρει σε πέρας στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπημένη θέση μεταξύ των πολλαπλών στόχων που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, απλώς θέλω να, να τοποθετηθώ για τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το επιχείρημα ότι το να αυξήσουμε την κεφαλογική τις κεφαλογικές απαιτήσει των τραπεζών θα μειώσει τη χρηματοδότηση προς την πραγματική αγορά. Είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε πιο συγκεκριμένα μέσα στα διάφορα μοντέλα τραπεζικής δραστηριότητας που έχουμε στις χώρες μας ακριβώς ποιο θα είναι το ποσοστό των δραστηριοτήτων τους που κατευθύνεται προ την χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με το ποσοστό του τζίρου τη που ασχολείται με την αγορά κεφαλαίων και με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. <clears throat> Γιατί το να έχουμε ένα τέτοιο επιχείρημα συλλήβδιν, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν οι διάφορες δραστηριότητες των τραπεζών για κάθε χώρα, ουσιαστικά είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι εύκολο με να το χρησιμοποιήσει κανείς, αλλά είναι επισφαλές, είναι επικίνδυνο. Γιατί παράλληλα ξέρουμε ότι οι υπερβολικοί κίνδυνοι και οι υπερβολικές απώλειες έχουν οδηγήσει στο να αναγκαστούν οι φορολογούμενοι να δώσουν τεράστια ποσά στις τράπεζες. Σύμφωνα με τον Ζουάο Μπαρόσο μιλάμε 4,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συνολική χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους προς τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον στη ζώνη του ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών. Αυτό είναι μια διαδικασία που είναι ακόμα εν εξελίξη. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι αποσύρονται όλα αυτά τα κονδύλια από την πραγματική οικονομία. Επομένω, μέσα στα πλαίσια αυτή τη αναζήτηση μια ισορροπία θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η εγκυρότητα αυτού του επιχειρήματο ότι με την αύξηση τη κεφαλογική επάρκεια των τραπεζών θα θυγεί η πραγματική οικονομία. Δεύτερο θέμα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην απολέσουμε τους στόχους που έχουμε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πολλοί συνάδελφοι αναφερθήκαν σε αυτό το θέμα. Πράγματι, με την πρωτοβουλία της Κομισιόν, η πρωτοβουλία αυτής της Κομισιόν μπορεί προς το παρόν να έχει τεθεί στο ψυγείο, να έχει αναφληθεί η εφαρμογή της, αλλά η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε μας οδηγούν κάθε φορά να απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από την πραγματικά ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της κρίσης των τραπεζών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε φυσικά έχουν μία σαφή θέση για τα ζητήματα αυτά. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέση της Κομισιόν ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικό της ταμείο διάσωσης τραπεζών και η κάθε χώρα έχει αναπτύξει το δικό της πλέγμα για να αντιμετωπιστεί το τραπεζικό πρόβλημα και παρά το γεγονός ότι οι κρίσεις αυτές έχουν οξυνθεί τον τελευταίο καιρό, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη μιας σαφούς προσπάθεια σύγκλησης των εθνικών λύσεων για την αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων. Γίνονται λοιπόν σε ασυνάρτητο επίπεδο οι προσπάθειες των κρατών μελών. Βλέπουμε σήμερα το πρόβλημα με την δέξια και βλέπουμε ότι ακόμα, σε ακόμα και σε χώρες που βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρώπης, στο κέντρο της Ευρώπης, δεν υπάρχουν <clears throat> επαρκείς μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν τραπεζικά προβλήματα. Ή λοιπόν θα πρέπει να επανέλθουμε στο να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη μέθοδο αντιμετώπισης των κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή θα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει όλο και μεγαλύτερη ανάμειξη και αλλη, αλληλορύπανση των τραπεζικών προβλημάτων και του, και του κρατικού χρέους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτά τα οποία ε, ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση πρωτοβουλία που ήμουν εγώ εισηγήτρια για τα θέματα αυτά. Ένα ακόμα σημείο, τρίτο σημείο, είναι απαραίτητο να έχουμε μια ισορροπία και μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων που ισχύουν στους διάφορους εθνικούς χώρους σε σχέση με τις διαφορετικές δραστηριότητες των τραπεζών, όπως το είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι. Πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση πιστοτικών ιδρυμάτων όπως αυτά που είναι τα ταμεία σύνταξη, τα συνταξιδοτικά ταμεία, Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης και σε μια πιο ουδέτερη αντιμετώπιση σε σχέση με το μειονοτικό κεφάλαιο που είναι σε πάρα πολλές τράπεζες σημαντικό. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά η ευελιξία αυτή δεν μπορεί να ε, να μας κάνει να ξεχάσουμε την ανάγκη να υπάρχει μια ενιαία ελάχιστη βάση που είναι απαραίτητη σε ένα ευρύ χώρο όπως είναι ο ευρωπαϊκός χώρος. Μια τελευταία παρατήρηση. Είναι απαραίτητο, όπως το είπε και κάποιος, να μην παραγνωρίσουμε την ύπαρξη της ε, σκιώδους τραπεζικής δραστηριότητας, του shadow banking. Όσο περισσότερο εμείς ρυθμίσουμε τον τραπεζικό τομέα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μεγαλύτερο θα είναι ο πειρασμό να δημιουργηθούν παράλληλε δομέ όπου μπορούν να συγκεντρωθούν υψηλοί συστημικοί κίνδυνοι. Γι' αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να παρατηρούμε την κατάσταση στο shadow banking και να μην παραγνωρίσουμε την ύπαρξή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε λιγότερο απαιτητικοί στη ρύθμιση και στην ενίσχυση της ευρωστίας των κανονικών τραπεζών. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, Σάρον, και ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο προηγουμένως. Ευχαριστώ, Σιλβί, στις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο γενικού τύπου παρατηρήσεις. Η πρώτη. Πιστεύω ότι πάνω σε αυτό το κείμενο αν και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Καρά, στον εισηγητή, δεν αμφισβητώ τις ικανότητές του, αλλά θα ξαναπέσουμε στο δίλημα που ζήσαμε σχετικά με το six-pack. Απ' τη μία δηλαδή καλούμεθα να νομοθετήσουμε για το μέλλον, αυτή τη στιγμή όμως το παρόν, η συγκυρία και η διαχείριση της κρίσης ε, μας απασχολεί πλήρως. Δεν είναι εύκολο. Ο Διώγος συμφωνεί μαζί μου. Και η Ελίζα επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει κανείς σωστά. Το μέλλον είναι αβέβαιο, συνάδελφοι. Δεν ξέρω πού θα βρισκόμαστε την επόμενη άνοιξη. Λυπάμαι ε, που δεν άκουσα κάποιους από τους συναδέλφους και βγήκα έξω γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν τρελαθεί για την δεξιά. Τι κάνουμε, συζητάμε για το μέλλον, για κανόνες που ίσως κάποτε εφαρμοστούν στα πλαίσια μιας κατάστασης για την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα και η οποία θα είναι χειρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε με τον εισηγητή, αλλά υπάρχει ένα θέμα τώρα. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν σχετικά με το Ταμείο Σταθεροποίησης και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί και για τα πιστοτικά ιδρύματα. Το δεύτερο το είπε η Ελίζα, δεν θα επιμείνω σε αυτό. Αυτό το οποίο όμως φοβάμαι και εγώ είναι ότι τις επόμενες, τις μέρες που θα έλθουν, θα δούμε να καταστρέφεται η εσωτερική χρηματαγορά γιατί δεν ακολουθήσαμε αυτά τα οποία εμείς είχαμε κάνει σαν προτάσεις και συστάσεις τότε με την ε, έκθεση πρωτοβουλίας ε, της Ελιζά, με τις προτάσεις Μαργκάλιο. Έχουμε να κάνουμε με κυβερνήσεις κρατών μελών που θα ανακεφαλοποιήσουν ε, μεμονωμένα τις τράπεζες γιατί υποτίθεται ότι έχουν βάρος σε μια χώρα, έχουν την έδρα σε μια χώρα καταστρέφοντας την διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Και όταν λένε το EBA δεν έχει πολλά μέσα, δεν έχει πολλά μέσα γιατί εμείς δεν του δώσαμε. Η εποπτεία θελήσαμε εμείς να είναι κάτι το πανευρωπαϊκό. Και στη Γερμανία υπάρχει ένας τέτοιος εκπρόσωπος εποπτικής αρχής που συνεχίζει να εργάζεται σε εθνικό επίπεδο ε, και ε, κοιτάει την αυλίτσα του, το οικοπεδάκι του και όχι προς τα έξω. Προφανώς, καλό είναι να σκεφτούμε υπό κανονικές συνθήκες το τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ίσως εδώ να λέω πράγματα που όλοι ξέρετε. Νομίζω όμως ότι το κοινοβούλιο μας έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι ένας από τους λίγους χώρους μαζί με την Κεντρική Τράπεζα ίσως, ίσως και την Επιτροπή, ε, στους οποίους προσπαθούμε να σκεφτούμε με ευρωπαϊκό τρόπο. Άκουσα αυτά που είπαν το Λίν. Καλό είναι να μπαίνει κανείς στη λογική του να λέει ότι πρέπει να είμαστε ουδέτεροι σε σχέση με τα εθνικά πρότυπα κτλ. Δεν ε, είναι κακά αυτά που λέει, αλλά το θέμα είναι να δούμε αν θα ευνοήσουμε τελικά την εσωτερική αγορά και όχι τη διαιώνιση εθνικών επιλογών, σεβαστών κατά τα άλλα, αλλά όχι χρήσιμων πλέον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια επιλογή, παρξιακή επιλογή σε σχέση με τη διαιώνιση της εσωτερικής αγοράς από τη μία ή τη διαιώνιση από την άλλη εθνικού τύπου οργανισμών οι οποίοι δεν επηρεάζουν θετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Νότμαρ για απαντήσεις. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια. Πράγματι οι καιροί είναι δύσκολοι και είναι σαφές ότι θα υπάρξουν μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν για να σταθεροποιηθούν οι αγορές. Έχουμε ξεφύγει λίγο από την κανονικότητα αν θέλετε. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την κατάσταση. Ήδη είχα πει και στους υπουργούς στο ανεπίσημο εκοφήν που έγινε στην Πολωνία στο οποίο αναφέρθηκα χθε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει το ψήφισμα για την κρίση να είναι τμήμα του πακέτου εποπτείας. Αυτό όμως δυστυχώς δεν έγινε δεκτό. Δεν έγιναν δεκτές όλες οι ιδέες μας. Αν είχε γίνει αυτό θα είχαμε κάτι σαν, στη διάθεσή μας σαν μέσο αντιμετώπισης του προβλήματος. Να υπενθυμίσω στα μέλη επίσης ότι έχουμε και άλλες νομοθετικές προτάσεις οι οποίες ε, περιμένουν. Ο κανονισμός σαν παράδειγμα που ε, ακαλύπτει τα ε, ταμεία που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νομισματικό τις εξειδικεύσεις, τις σκιώδεις πιστοτικές δραστηριότητες, γιατί αυτές οι σκιώδεις τράπεζες ουσιαστικά δεν είναι κανονικές τράπεζες, δεν είναι πλήρεις τράπεζες και είναι σαφές ότι ε, θέλουμε εμείς να υπάρχει διαφάνεια και σε αυτές τις δραστηριότητες, θέλουμε να υπάρξει, ε, υπάρξουν καλά στοιχεία θετικά στοιχεία, αν και ίσως σε αυτή τη φάση δεν είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Ότμαρ τώρα, θέλεις το λόγο να δώσεις κάποιες απαντήσεις ή να σχολιάσεις κλείνοντας τη συζήτηση. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για το πλήθος τοποθετήσεων και αντιδράσεων. Η κάθε μία τοποθέτηση έδειξε όμως με πόση σοβαρότητα η παρούσα Επιτροπή αντιμετωπίζει το θέμα και με πόση ευαισθησία. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για τα καλά σας λόγια, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου. Και να μπορέσω λοιπόν να ανταποκριθώ σε αυτό και να σας δικαιώσω χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Και για τη συνέχιση αυτού του ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου θα ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικά σχόλια εκ των προτέρων. Πολλοί από εσά εκφραστήκατε υπέρ της ισορροπίας και ε, της ε, αναλογικότητας. Αλλά η ισορροπία δεν είναι το να ικανοποιούνται όλες οι ειδικέ επιθυμίες. Ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής δεν χρειάζεται απαραίτητο να είναι πάντα ισορροπημένος. Και η ε, προσοχή και η συμπερίληψη όλων των ειδικών μεμονωμένων συμφερόντων, κρατικών ή ατομικών, δεν θα πρέπει να ε, είναι κάτι που να οδηγεί σε ισορροπία. Θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πού στοχεύουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους σε σχέση με αυτό που είπε η Σιλβί Γκουλάρ. Η εσωτερική αγορά και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς είναι στόχος, μάλιστα απαντώ. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς και όχι των μεμονωμένων ε, κρατικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρέπει να ξαναπώ το εξή. Το αν θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας δεν έχει πάντα να κάνει με την οδηγία. Μπορεί να έχει σχέση με την οδηγία ε, γιατί υπάρχει υπάρχει δύο πόρων, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα υπάρξει πρόβλημα ε, Και στη Βασιλεία 2 μιλήσαμε για την πιστοληπτική ικανότητα ε, των επιχειρήσεων. Το θέμα είναι πώς θα ρυθμίσουμε αυτό το θέμα για να μην υπάρξει αυτή η πιστοτική στενοπός ή να μην ε, ακριβίνουν οι χορηγήσεις για να περιορίσουμε όσο γίνεται αυτό το κίνδυνο. Αλλά να τον αποκλείσουμε δεν μπορούμε ποτέ. Πολλοί από σας μιλήσατε για το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων. Αυτό μας ενδιαφέρει πραγματικά μόνο το ποσοστό. Αλλά τι αξιολογούμε εμείς, τι ορίζουμε ως ίδιο κεφάλαιο. Γιατί είναι και ένα ζήτημα ορισμού ιδίων πόρων, ιδίων κεφαλαίων. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει μια νομική ουδετερότητα και να είναι αρχή αυτή. Σήμερα έχουμε την εξή κατάσταση. Μας λένε κάποιες επιχειρήσεις και μεγάλοι όμιλοι ότι αυτή η ρύθμιση ε, τους οδηγεί στους υπολογισμούς τους στο 1 τρίτο είδη του υπάρχοντος κεφαλαίου πριν ε, καν έχουν τζίρο ενός ευρώ λόγω και των μικρών ε, ε, συμμετοχών, των μικρομετόχων το μερίδιο δηλαδή της ε, ε, ε, το θέμα της στάθμισης του κινδύνου και άλλα ζητήματα ε, μπαίνουν και έχουν σημασία και όχι μόνο το ποσοστό για να ορίσουμε τι εστί ίδιο κεφάλαιο. Και βέβαια, βέβαια θέλουμε ευελιξία, αλλά η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει και σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αυτό τον καιρό συζητούμε ε, τα θέματα κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, τα buffers, που είναι σημαντικά και πού οδηγεί αυτό. Αυτή τη στιγμή και οι εθνικές εποπτικές αρχές της έδρας της εταιρείας απαιτούν περισσότερα ίδια κεφάλαια από τη τράπεζα αυτή λόγω της εξωτερικής της δραστηριότητας από ό,τι απαιτούν από τράπεζες που δραστηριοποιούνται μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή και αυτό είναι μια επιπλέον ε, απέτηση ιδίου κεφαλαίου. Έτσι ώστε αυτό να οδηγεί ενδεχομένως ε, σε ε, υπερβολική επιβάρυνση, άρα και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ναι λοιπόν, στην ευελιξία αλλά πού είναι το σύνορο και η διαχωριστική γραμμή με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά και με μεγάλη ευαισθησία. Δεν είναι θέμα ορισμών και όρων. Όλοι συμφωνούμε με την έννοια της ευελιξίας και με τις συμπεριλήψεις και τις προσοχής, ό,τι θέλετε. Όλοι ικανοποιούμαστε και συμφωνούμε μέσως. Βέβαια, όταν έρχεται στο συγκεκριμένο τι σημαίνει αυτό σε κάθε ρύθμιση, για να έρθω και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την ΕΜΠΑ. Βεβαίως χρειαζόμαστε υποστήριξη. Ο Μάριο Νάβα έκανε μια πολύ ωραία ε, παρουσίαση, μας ενημέρωσε. Πριν από μια-δύο εβδομάδες πολλοί ήσασταν εδώ, αλλά και περισσότεροι ήταν οι βοηθοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι όταν απευθύνεται στην αρχή αυτή χρειάζονται πολύ περισσότεροι υπάλληλοι. 8 ε, ακούσαμε, τώρα ε, ενδεχομένως να είναι και 10 με όλες αυτές τις αποστολές που τις αναθέτουμε. Και θα πρέπει να το λύσουμε και το οικονομικό και το προσωπικό, αλλιώς θα υπάρξει διάσταση ανάμεσα στις συζητήσεις που κάνουν εκεί και τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς και θα έχουμε και ε, προβλήματα χρονικά που δεν θα συμπίπτουν οι συζητήσει μας και θα πρέπει να κάνουν και μια διάκριση μεταξύ των τριών ενωτήτων που αναλαμβάνει τώρα η αρχή ότι είναι σύσταση τι είναι άμεση εφαρμογή και τι είναι γενικά ανάλυση και θεωρία. Αλλά εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να ε, μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τι είναι αυτές οι 153 αναθέσεις, ε, εφαρμοστικές πράξεις. Χρειάζεται ένας παράλληλος διάλογος με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τράπεζων και ε, με την δική μας Επιτροπή ε, στην εκπόνηση των νομοθετικών κειμένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα πρέπει να, να πληρωθούν οι προϋποθέσεις και κάλυψης προσωπικού. Περί αυτού πρόκειται. Και θα το ε, αντιμετωπίσουμε και θα ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά παρακαλώ να πρετανεύσει το ίδιο πνεύμα όπως και σήμερα, αλλά με μεγαλύτερη ευάθυνση και μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Και μετά να γίνεται διμερός η συζήτηση. Γιατί με το να δηλώνουμε απλώς ευελιξία δείχνουμε μεγάλη ε, ελπίδα και με την ισορροπία, πολύ ωραία αυτά, αλλά συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό απέναντι στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η βάση για τη δική μας εργασία είναι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάνω από αυτή, μάλλον πλαίσιο αυτή είναι η Συμφωνία της Βασιλείας και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με όλα αυτά που λέμε εμείς είναι βελτίωση και ευάθυνση, ωραία, και έχουμε και το G20 από πάνω. Δηλαδή, ε, είναι τρία τα επίπεδα στα οποία έχουμε ε, δεσμευτεί. Και θα πρέπει να δούμε πόσο μεγάλο είναι το περιθώριο ελιγμών. Γιατί όλα αυτά ε, είναι ένα γρανάζι το οποίο συνδέεται. Και εμείς κινούμε από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθετική μας εργασία, αλλά στο θέμα της εφαρμογής των δικών μας ε, απαιτήσεων και απέναντι στους Αμερικανούς για να έχουμε ίσους όρους παιχνιδιού διεθνώς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις αποφάσεις της ε, Βασιλείας και των G20. Θα πρέπει να γίνει αυτό το τμήμα της δικής μας επιχειρηματολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Ας ανασκουμποθούμε λοιπόν και Ας διατηρήσουμε μέχρι την ψηφοφορία του χρόνου την εμπιστοσύνη που σήμερα έγινε τόσο αισθητή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες Καθίστε, η έκθεση θα εξεταστεί στις 23 Ιανουαρίου το σχέδιο έκθεσης και ελπίζουμε ότι ο Όθμαρ έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Η προτινόμενη Προθεσμία για τροπολογίες 27 Φεβρουαρίου, 20 Μαρτίου θα εξεταστούν οι τροπολογίες και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 25 Απριλίου, Ολομέλεια, η 1η του Ιουνίου 2012, αν θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το τωρινό χρονοδιάγραμμα και θα έχουμε βέβαια και ακροάσεις οι οποίες θα μας δώσουν περαιτέρω πληροφορίες πριν <clears throat> φτάσουμε στην τελική μορφή του σχεδίου έκθεσης. Μπορούμε τώρα λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη που είναι το 9, η μεταρρύθμιση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κρατικές ενισχύσεις σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Αν κάποιοι θέλουν να φύγουν, ίσως πρέπει να κάνουμε δύο λεπτά διακοπή για να μην προσπαθεί ο κύριος Σίμων να μιλήσει πάνω από την γενική φασαρία. Όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν τώρα παρακαλώ ηρέμος και ησύχος. So those, those leaving, please hurry up. Παρακαλώ όσοι φεύγετε ησυχία για να συνεχίσουμε. Right. I'm going to ask those who are... Θα ζητήσω λοιπόν από όλους ε, όσοι έμειναν στην αίθουσα να καθίσουν παρακαλώ. Then I can judge who's here and who's going. Okay, is everybody who's departing departed? Okay, right. So we're now going to, I'm going to give the floor. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο για μια παρουσίαση ε, των τροπολογιών, Πίτα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την επικοδομητική σας συμβολή. Υπήρξαν πολλές τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν είναι πιστεύω προφανές ότι θα πρέπει να έχουμε συμβαστικές ε, λύσεις για πάρα πολλά σημεία. Υπάρχουν βέβαια μερικά επίμαχα σημεία τα οποία εκφράζονται από τις τροπολογίες και τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ θέλω να σταθώ τώρα σε τρία από αυτά τα σημεία. Πρώτα απ' όλα το άρθρο 14, το θέμα του νομικού πλαισίου. Δεύτερον, των κανόνων de minimis κατά περιοχή και το τρίτο είναι το επίμαχο σημείο της αποτελεσματικότητας. Έχουμε το κείμενο της Κομισιόν για τις, ε, τους νέους κανόνες επιδοτήσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Έχουμε την πρόταση λοιπόν της Κομισιόν, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά θέλω να έρθω καταρχήν στο άρθρο 14 και το νομικό πλαίσιο. Είναι σαφές ότι η πρότασή μας να έχουμε ένα οριζόντιο πλαίσιο για τις επιδοτήσεις ήταν μια γενική απέτηση, αλλά οι συζητήσει οι οποίε έγιναν τον προηγούμενο χρόνο και οι συζητήσεις που έγιναν στο, στην Επιτροπή μας το έχουν καταδείξει. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσω ότι εμείς ως Σοσιαλδημοκράτε, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο επί τη βάση του άρθρου 14 αυτές τις επιδοτήσεις, γιατί αυτό μπορεί να έχει αποτελέσματα αρνητικά στον ανταγωνισμό. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 14. Η Κομισιόν έχει την έννοια για τις υπηρεσίες αυτές, υπηρεσίες που έχουν εταιρείες, που έχουν ε, δημόσιες λειτουργίες, κρατικές υπηρεσίες κτλ. Εδώ τι το πρώτο ερώτημα προς τους συναδέλφους και ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές. Συμφωνείτε ότι η απαρίθμηση της Κομισιόν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφαλή δικαίου, η απαρίθμηση δηλαδή των φορέων που είναι γενικού οικονομικού συμφέροντος. Αν λοιπόν κάποιο ο οποίο δεν ανταποκρίνεται, ένα που αν δεν ανταποκρίνεται σε, αυτούς, σε αυτά τα κριτήρια τη Κομισιόν, δεν μπορεί να την χάνει επιδοτήσεων. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια σαφήνεια. Επίση, ο Επίτροπο Αλμούνια την Παρασκευή ε, αναφέρθηκε και στο πλαίσιο ποιότητος και το πρωτόκολλο 64 στα πλαίσια του άρθρου 14. 26 Και το, το ερώτημα είναι μήπως θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερα ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή προτού η Κομισιόν δώσει τη δική της ερμηνεία να εκφράσουμε τη θέση μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι κανόνες de σε συγκεκριμένους τομείς. <clears throat> Μέχρι το 2013 θα παραμείνει η υφιστάμενη ρύθμιση de minimis και θα ανανεωθεί στο τέλος του 2013. Αλλά έχουμε δύο συγκεκριμένες περιοχές. Καταρχήν, για δήμους και κοινότητες οι οποίες έχουν μια κοινοτική αρχή η οποία ε, δεν μπορεί πάντα να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές για τις τοπικές, ε, για τις επιδοτήσεις αυτές και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος γενικά στην περίπτωση αυτή δεν προξενούν κάποιο κίνδυνο στρέβλωση τη εσωτερική αγορά. Δεύτερον, κοινωνικές παροχές υπηρεσιών οι οποίες <clears throat> δεν θα επηρεάσουν την αγορά και το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Θέλουμε ιδιαίτερα να έχουμε κανόνες δε για τους μικρότερους δήμους και κοινότητες. Η Κομισιόν έχει προτείνει μια πρόταση στο επίπεδο αυτό. Όταν πρόκειται για λιγότερο 150.000 ευρώ τον χρόνο για δήμους κάτω των 10.000 ε, πολιτών, κατοίκων και για επιχειρήσεις με τζίρο κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά θα ήθελα στον τομέα να υπενθυμίσω το εξή. Εγώ θεωρούσα ότι ιδίω για τι μικρέ διοικητικέ αρχέ να υπάρχουν εξαιρέσει. Αλλά μπορεί να υπάρξει και για λόγους επηρεασμού της εσωτερικής αγοράς ένα όριο σε σχέση με το επίπεδο της επιδότησης. Η Κομισιόν έχει προτείνει το όριο αυτό των 10.000 κατοίκων για να περιληφθούν αυτές οι, οι δήμοι και, ο κύριος Σαλμούνια την τελευταία στιγμή έχει πει ότι θα μπορούσε να δεχτεί αυτήν την ε, λύση. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας, ποιες είναι οι προτάσεις σας. Είναι ανοιχτά ακόμα είναι ανοιχτή ακόμα η θέση μας για τα κριτήρια σε σχέση με την αντίδραση που πρέπει να έχουμε στην πρόταση της Κομισιόν. Υπήρξε μια πρόταση από τον Οκρανή που είχε προτείνει ένα χρόνο ένα χρονικό διάστημα τριών ετών για να εξισωθούν οι επιδοτήσεις αυτές. Τώρα, για την παροχή υπηρεσιών. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική άποψη ότι δυστυχώς η Κομισιόν δεν έχει κάνει κανένα, καμία ρύθμιση ντεμίνιμης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να καλυφθεί όμως η μεγάλη κοινωνική ανάγκη που υπάρχει και να απελευθερωθούν πραγματικά τα νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες στέγασης από την ανάγκη κοινοποίησης στην Κομισιόν σε περίπτωση μιας επιδότησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν ότι αυτό θα ήταν μια πραγματικά μεγάλη ελάφρυνση για τις υπηρεσίες αυτές, αλλά από μόνο του αυτό δεν υπάρχει Τέλος, αναφέρθηκε και το θέμα της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. <clears throat> Στο κείμενο της Κομισιόν, σε σχέση με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιδοτήσεις, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες παροχές υπηρεσιών θα πρέπει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν και κριτήρια ε, αποδοτικότητος για να μπορέσουν να γίνονται αυτές οι επιδοτήσεις με τρόπο ο οποίος είναι συμβατός προς την εσωτερική αγορά. Προφανώς λόγω της κατάστασης του προπολογισμού των κρατών μελών, τα κίνητρα αυτά είναι κάτι το επενετό, κάτι το οποίο θα θέλαμε όλοι. Αλλά όπως τονίστηκε ήδη στην Επιτροπή μας στο παρελθόν, στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει κανένα, καμία νομική βάση για αυτή την πρόταση που κάνει η Κομισιόν για τα κίνητρα αυτά. Για τις ε, τροπολογίες τώρα, ε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν σε επίπεδο εθνικό και όχι σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αλλιώς θα χρειαστεί ίσως ένας κανονισμός ο οποίος να θεσπίσει τα θέματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την παροχή κινήτρων. Το άρθρο 14 λοιπόν πρέπει να είναι η βάση για τα θέματα αυτά. Η Κομισιόν παραγνωρίζει ακόμα και την αρχή της επικουρικότητος και τους κανόνες της ευρωπαϊκής ε, των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Δεν μπορώ λοιπόν να μην κάνω μια σαφή μηνία προς την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας για τα θέματα αυτά των τροπολογιών, ώστε να μπορέσει αυτή η έκθεση, χάρη σε επικοδομητικές συμβιβαστικές λύσεις που θα μπορέσουμε να σφυριλατήσουμε όλοι μαζί, να έχει το αποτέλεσμα που προσδοκούμε. Ευχαριστώ και εγώ. η Σοφίντβελτ, αλλά πρώτα Χακμακ, Σκίνα για τους συντηρητικούς ή την υπάρχει κάποιος Η κυρία Ισαγιά, η κυρία Οκονή ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί υπάρχει μια σημαντική ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα παρουσιάσω λοιπόν τις απόψεις της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμφωνεί με, το, με τη βάση αυτής της μεταρρύθμισης που ε, εδράζεται θα έλεγα στη βασική αρχή της απλοποίησης. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να συντάσσουμε τις τροπολογίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το νέο σχέδιό της, το πλήρες κείμενο, δύο ανακοινώσεις, ένας κατάλογος ε, εξαιρέσεων και ένας κανονισμός de minimis. Το πρόβλημα είναι ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αν θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας αυτό το νέο κείμενο, στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τον εισηγητή. Ίσως το συμβιβαστικό κείμενο να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις ε, ιδέες αυτές. Το θέμα που τίθεται με το κείμενο αυτό είναι αν οι καινούργιοι κανόνες εξυπηρετούν το στόχο της απλοποίησης. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω τρία θέματα. Πρώτον, να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες και μετά να αναφερθώ στους κανονισμούς de Κάποιες διευκρινήσεις εννοιών είναι κάτι το απροαπαιτούμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι προσπαθεί να ορίσει σωστότερα προσπαθώντας ε, να εντάξει σε νομικό κείμενο της, ε, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι εννοεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναφέρεται σε μια τέτοια υπηρεσία σαν γνήσια υπηρεσία καθολικού συμφέροντος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και οι εξηγήσει τις οποίες ε, έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σελίδα 7 και 8 της ανακοίνωσής της ε, δεν επαρκούν και δεν είναι κατανοητές. Αν δεν καταλαβαίνουμε εμείς το κείμενο αυτό διαρωτώ με πως ο υπόλοιπος κόσμος που τον ενδιαφέρει το θέμα αυτό θα μπορούσε να ασχοληθεί. Τώρα για τους κανονισμούς de ε, Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση του επίπεδου de για τη διασφάλιση κοινωνικών υπηρεσιών, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που δεν επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές. Το όριο το οποίο θέτει είναι το 10.000 κάτοικοι. Αυτό δεν είναι κατάλληλο. Βέβαια από τη μία χώρα σε άλλη υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές στις πληθυσμιακές ε, ε, συγκεντρώσεις και εδώ είναι κάτι που οι χώρες μπορούν ίσως να βοηθήσουν. Το μόνο, ε, το μόνο θα έλεγα κατανοητό είναι το επίπεδο, το ύψος της δημόσιας επιδότησης. Θα πρέπει να εμείνουμε λοιπόν στην μέθοδο ε, εξέτασης των στοιχείων τα οποία παρέχονται και της τεκμηρίωσης των στοιχείων. Για τις εξαιρέσεις και εδώ η απλοποίηση είναι καλοδεχούμενη. Η απλοποίηση όμως δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της διαφάνειας. θα πρέπει στα πλαίσια της εντολής που έχουν ε, τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να δώσουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, αλλά να μην υπάρχουν υπερβολικές αποζημιώσεις, να μην υπάρχουν υπερκαλύψεις του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την απαιτούμενη νομική ασφάλεια mm και θα πρέπει ακριβώς όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει καλύτερα το τι εννοεί α, με βασικές ανάγκες. Συμφωνούμε επί της αρχής. Υπάρχουν όμως όπως είπα αρκετά στοιχεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Ελπίζουμε οι συμβιβαστικές τροπολογίες να μας επιτρέψουν να το κάνουμε. Θα ήθελα να επιθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ότι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη στα θέματα του ανταγωνισμού. Αλλά παρόλα αυτά νομίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι χρήσιμο για τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες είναι τόσο κοντά στις ανάγκες του πληθυσμού σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ. Η Σόφη Ινβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. To ε, Χαίρομαι που ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη ιδεολογίας. Αυτό προσπαθούμε τόσο καιρό να κάνουμε, χρόνια ολόκληρα. Αν κοιτάξετε τη συνθήκη, όλα τα αντίστοιχα άρθρα της συνθήκης είναι τελείως ουδέτερα. Δεν προκρίνουν κανένα ε, μοντέλο και αφήνουν τα κράτη-μέλη να οργανώσουν όπως θέλουν αυτές τις υπηρεσίες ε, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών τους. Αυτό θα πρέπει να ισχύει άλλωστε. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολύ επιφυλακτική, προσεκτική, ουδέτερη, καθόλου ιδεολογική προσέγγιση. Ο Επίτροπος Αλμούνια προσπαθεί σαφέστατα να φέρει λύσεις πολύ στοχευμένες και κομμένες και ραμμένες στα μέτρα αναλόγως. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να έχουμε εγκάρσιες ε, ε, εξαιρέσεις, δε μήνυμη ή πλαίσια διάφορα νομοθετικά. Εκεί μπαίνουμε στην ιδεολογία. Οποιαδήποτε γενική αντιμετώπιση, οριζόντια μέτρα δεν δικαιολογούνται να καλύπτουν. Έχω πολλά ερωτηματικά. Το 2005 συζητούσαμε το πακέτο Monty Cruz το ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ξεπέρασε. Ήταν πολύ πιο γενναιόδορη στις ε, οριζόντιες και εγκάσεις, ρυθμίσεις που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Δεν έχω ενθουσιαστεί απαραίτητο από ε, Όσες φωνές ζητούν να διευρυνθούν αυτά τα μέτρα χωρίς λεπτομερή αιτιολόγηση και δικαιολόγηση. Κοίταξα τις τροπολογίες. Τρία είναι τα ζητήματα που θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα. Πρώτον, προτάσεις για νομοθετικό πλαίσιο για το γενικό οικονομικό συμφέρον. έκαθεν ήμασταν αντίθετοι, ποτέ δεν υπήρχε πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ομάδα μου δεν θα αλλάξει στάση για τους λόγους που μόλις σας εξέθεσε αν θέλουμε ε, διευκρίνηση και απλούστευση, εντάξει, αλλά εάν δεχτούμε ότι τα κράτη-μέλη θα ορίζουν μόνα τους πώς θα οργανώνουν αυτές τις υπηρεσίες και πώς θα χρηματοδοτούνται, με αυτό δεν χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο. Είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δεύτερον, για τον κανόνα ντεμίνιμις και πάλι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εδώ. Συμφωνούμε με το στόχο της απλούστευσης και ε, της κατάργησης της περιττής γραφειοκρατίας, αλλά θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να μελετήσουμε τα κριτήρια. Τώρα αυτό το γενικό κριτήριο για το μέγεθος του Δήμου ή της κοινότητας μπορεί να φαίνεται απλό και ε, εύκολο, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Να δούμε ποιο θα είναι ο αντίκτυπος. Και τέλο, γίνεται ειδική αναφορά στην έκθεση ε, για ε, τις Ολλανδικές Ενώσεις ε, στέγη, Στέγασης. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κατονομάζουμε κάποιους και να τους στιγματίζουμε. Αλλά η χώρα μου βέβαια δεν αναφέρεται ρητά, αλλά αυτά που λέγει η έκθεση είναι ανακριβή. Οι ενώσεις αυτές ε, λέει, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη για εμπορικέ δραστηριότητες σύμφωνα με μια απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι τελείως ανακριβές και λάθος. Αν γίνεται λόγο λοιπόν για τις ε, κοινωνικές κατοικίες ε, στις κάτω χώρε να σας δώσω ό,τι στοιχεία θέλετε, αλλά αυτά που λέγει αυτή τη στιγμή η έκθεση είναι τελείω ανακριβή και ξέρω και από πού προέρχονται και διαφωνώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πασκάλ. Oui, moi j'ai <coughs> toujours Με μεγάλη χαρά σα υπενθυμίζω πάντα ότι συζητούμε αυτή την ρύθμιση για τις κρατικές επιδοτήσεις, ενώ ίσως σε μερικές ε, μέρες θα, οι δημόσιες αρχές θα κάνουν μια ένεση μερικών δισεκατομμύριων ή δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στο τραπεζικό σύστημα χωρίς να ενοχληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, στρέβλωση ανταγωνισμού. Έχουμε ανανέωσει λοιπόν αυτές τις μαζικές εξαιρέσει για τον τραπεζικό τομέα. Είναι πραγματικά υπερβολικό και παράδοξο να κοιτάμε για μερικές ε, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τους κανόνες δε για τους Δήμους και τις κοινότητες όταν δίνουμε τεράστια <clears throat> ποσά σε τραπεζικά ιδρύματα. Ίσως θα πρέπει να έχουμε και μία μια έννοια ισορροπίας, μια έννοια της σωστής διάστασης σε ό,τι αφορά τα θέματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί από τον Πίτερ Ζήμον και έχω το ίδιο ερώτημα, όπως και η συνάδελφός μου του ΕΛΚ. Πώς ακριβώς θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε το νέο κείμενο της Κομισιόν στις ε, τροπολογίες μας, γιατί έχει δημοσιευτεί μετά από την κατάθεση των πρώτων μας τροπολογιών το κείμενο, το νέο κείμενο της Κομισιόν. Πώς μπορούμε λοιπόν να τροποποιήσουμε τις τροπολογίες που έχουμε θέσει και επίσης ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν αφού είναι παρόν. Πώς προβλέπει η Κομισιόν να ενσωματώσει τη γνωμοδότηση του, την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εργασία που θα λάβει η χώρα στην Κομισιόν. Ξέρω ότι ο καθένα έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα και του δικού του περιορισμού, αλλά το γεγονό ότι έχει παρουσιαστεί επίσημα το κείμενο τη Κομισιόν μετά από την ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντίστοιχη έκθεση, <clears throat> αυτό δεν διευκολύνει την, τον διάλογο μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και θα μπορούσε να είναι και κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε δυσαρέσκεια των κοινοβουλευτικών. Δεν θέλω τώρα να επιλήψω την ευθύνη στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα ήθελα όμως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να μας πει πώς θα λάβει η Κομισιόν υπόψη την ε, θέση και τη γνώμη του Κοινοβουλίου στη διαδικασία η οποία ξεκινά τις επόμενες ε, ημέρες και εβδομάδες. Επίσης, για το όριο των 10.000 κατοίκων, νομίζω ότι όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι εύστοχο αυτό το κατόφλι. Εγώ βρίσκομαι στο ζω στο Παρίσι, όλες οι πόλεις, οι, οι συνοικίες και τα προάστια τα οποία είναι μειονεκτικά γύρω από το Παρίσι έχουν πληθυσμό πολύ περισσότερο από 10.000, δηλαδή μπορούμε να έχουμε περιοχές όπου δεν υπάρχει και ιδιαίτερο οικονομικό συμφέρον για μια εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία να παρέμβει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οι 10.000 πρέπει να είναι όριο. Υπάρχουν περιοχές γύρω από το Παρίσι που έχουν πολύ περισσότερο πληθυσμό και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα στρεβλώσει το εμπόριο για την ασφάλεια δικαίου και το άρθρο 14. Εγώ θα ήθελα επίση το ΕΛΚ <clears throat> να σκεφτεί καλύτερα, όχι ιδεολογικά, αλλά περισσότερο για το πώς θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η νομική ασφάλεια για τη χρήση του άρθρου 14. Γιατί αν κατάλαβα αυτά που είπε η βουλευτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλετε να υπάρχει μια σαφήνεια για την έννοια αυτή, αλλά παραμένοντας μέσα στην επικουρικότητα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια ιδέα, ότι πρέπει να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο επικουρικότητας, αλλά η επικουρικότητα μπορεί να, ισχύσει μονάχα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου. Από δημοκρατική έποψη λοιπόν δεν μπορούμε να φανταστούμε ο καθορισμός των ενιών του γενικού οικονομικού συμφέροντος και των εξαιρέσεων, όλα αυτά πρέπει <clears throat> να γίνουν με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο για το οποίο θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι η θέση της Κομισιόν επί της ουσίας είναι πολύ λιγότερο απομεμακρυσμένη από αυτά που πιστεύω εγώ, από ότι από αυτά που θα προέλθουν ίσως σε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ από τη δική μου πολιτική θέση ίσως θα θεωρούσα ότι θα ήταν καλύτερο να μην υπερασπιστούμε το άρθρο 14, αλλά από δημοκρατική έποψη είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διευκρινίσουμε θέματα που είναι τόσο σημαντικά για τους πολίτες και την καθημερινή του ζωή και όχι να αφήσουμε την Κομισιόν να παίρνει αποφάσεις μόνη της. Δεν είναι ότι δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση Κομισιόν, αλλά δεν είναι επαρκής για να πάρει τέτοιου είδου αποφάσει. Ένα τελευταίο ερώτημα και για τον Πέτερ Ζήμον και για την Κομισιόν. Είναι το θέμα των εξαιρέσεων. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στην πρόθεση της Κομισιόν. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο, κανον, ο κατάλογος είναι εξαντλητικός ή όχι Νομίζω ότι στο αγγλικό κείμενο εμφανίζεται σαν εξαντλητικό, στο γαλλικό κείμενο δεν εμφανίζεται σαν εξαντλητικό. Αυτό όμω είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνουμε, να ξέρουμε αν είναι εξαντλητικό ο κατάλογο των εξαιρέσεων ή όχι. Και θα ήθελα ο Πέτερ να μα εξηγήσει ποια είναι η δική του αντιμετώπιση, αν είναι ο κατάλογο πλήρη ή αφήνει περιθώριο και σε άλλε εξαιρέσει. <coughs> Γκούνερ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να ισορροπήσουμε από τη μία την επικουρικότητα και το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς από την άλλη. Βλέπουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν βάση εκκίνησης και για το θέμα αυτών, αυτής της μορφής των υπηρεσιών που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα από τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης σήμερα, όταν μιλάμε για το χρέος, είναι η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης. Και όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι οφείλεται εν μέρη στο ότι δεν ανοίξαμε τις εσωτερικές αγορές για νέες υπηρεσίες και χρησιμοποιήθηκε και η μεταφορά για τα τελεκόμ επανειλημμένα. Δεν θα μείνω σε αυτό. Πάντως νομίζω ότι περισσότεροι από εμά θεωρούν ότι τα πράγματα βελτιώνονται από τότε που οι εταιρείε Telecom ε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν μέσα σε ανταγωνισμό και δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει επιλογές. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους έχει σημασία ο ανταγωνισμός. Βέβαια όσο πιο εγγύς είναι η παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας προς τον πολίτη τόσο πιο σημαντικό είναι να είναι υψηλή ποιότητα, όσο υψηλότερη ποιότητα γίνεται και να βίβεται η υπηρεσία αυτή με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το αντίθετο είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ισορροπούμε λοιπόν από τη μία την επικουρικότητα με την εσωτερική αγορά. Αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε και γι' αυτό δεν χρειάζεται εδώ μια κάποια συνολικά οριζόντια νομοθετική απόφαση. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε το ότι οι υπηρεσίες αυτές οικονομικού συμφέροντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν άλοθη για την έλλειψη του ανταγωνισμού ή για την προάσπιση μονοπωλιακών καταστάσεων. Η σημαντική ισορροπία την οποία θα ήθελα οι συγητές να πετύχουν θα έλεγα, να μην αγνοήσουν τουλάχιστον, είναι η διαφορά ανάμεσα στη δημόσια από τη μία χρηματοδότηση κάποιων υπηρεσιών και από την άλλη την βοήθεια στις επιχειρήσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στα δύο, γιατί πάρα πολλά χρήματα τα οποία δίδονται έχουν σαν στόχο την χρηματοδότηση και την επιδότηση των δημοσίων υπηρεσιών και όχι τόσο των ίδιων των υπηρεσιών, της παροχής τους δηλαδή. Ξέρω τι γίνεται με την κοινωνική κατοικία στην Ολλανδία σαν παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να βελτιωθούν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν να, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι ζουν στα πλαίσια της λεγόμενης κοινωνικής κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν ανάγκες βελτίωσης της κατοικίας τους ακόμα και εκτός επιδοτουμένων κατοικιών. Λοιπόν, αν ακολουθήσουμε μία θα έλεγα γραμμή χωρίς να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα θα χειροτερεύσουμε την κατάσταση και βοηθάμε κάποιες ε, υπηρεσίες ε, οι οποίες δεν είναι και τόσο θετικές απέναντι στην ιδέα της εξυπηρέτησης ε, των αναγκών του καταναλωτή. Κάτι το οποίο είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Για να μην μακρηγορώ, θα ζητήσω τον, από τον εισηγητή όταν προχωρήσει στις συμβιβαστικές προτάσεις να μην σταθεί απέναντί τους με ιδεολογικό τρόπο και το είπε άλλωστε αυτό. Όταν κανείς προφεί ιδεολογικές απόψεις ε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις δομές του παρελθόντος αλλά τις υπηρεσίες του μέλλοντος προς τον καταναλωτή. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο. Και στα πλαίσια αυτής της διαφοράς υπάρχει ανάγκη επίσης σεβασμού της επικουρικότητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό όμω δεν είναι άλοθη για αναποτελεσματικότητα, μονοπόλια και μειωμένου ρυθμού ανάπτυξης. Ο στόχο μα πρέπει να είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Πίτερ Σκίνα like to think that the rapporteur has certainly got and has expressed a balanced view. Πράγματι άκουσα πολύ θετικέ ιδέε και χαίρομαι που ο Πίτερ Ζήμων είναι... Χαίρομαι που ο Πίτερ Ζήμων είναι ο εισηγητής σε αυτή την έκθεση. Έχει ενδιαφέρον να ακούει κανείς ότι υπάρχει και το θέμα της ιδεολογίας που μας επηρεάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα δεν είναι να έχουμε ιδεολογικές αντιλήψεις, το θέμα είναι να μην έχουμε ιδεολογικές ακρότητες οι οποίες να επηρεάζουν ακριβώς αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να είναι, δηλαδή η τέλεια αγορά. Δεν υπάρχει η τέλεια αγορά, δεν υπάρχει μια απόλυτα ομοιογενής αγοράς. Αν θέλει κανείς να σταθεί ιδεολογικά πάνω σε ορισμένα προβλήματα προς τη μία κατεύθυνση δεν μπορεί να αποκλείσει την ιδεολογία που προέρχεται από μία άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Αν θέλουμε να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την παροχή μιας υπηρεσίας προς την κοινωνία είναι σαφές ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σωστά πιστεύω στο κοινωνικό αγαθό, είναι κάτι το οποίο παρέχει σε μια ειρηνευτική δύναμη, στο στρατό ή στις υπηρεσίες υγείας. Υπάρχουν ανάγκες προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα μονολυθικά θεσμικά όργανα τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά σε ορισμένες χώρες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρέπει να βρούμε ένα έξυπνο τρόπο για να μπορέσουμε είτε να διατηρήσουμε ε, μια δομή υπηρεσιών είτε να δημιουργήσουμε μια νέα δομή υπηρεσιών για να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να γίνουμε Χονκ εδώ που είναι η αγαπημένη περιοχή του Μίλτον Φρίντμαν στον κόσμο, όπου όλα γίνονται με βάση τον χαμηλότερο δυνατό παρανομαστή, κοινό παρανομαστή. Ε, μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα εδώ, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει πάρα πολύ στον τομέα αυτό της απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Αυτό ξεκίνησε με τους νεοφιλελευθέρους, δεν ξέρω αν είναι κάποιος συντηρητικός από εδώ, που δεν πιστεύουμε οι περισσότεροι από εμά. Εκείνη την εποχή πίστευαν ότι ήταν απαραίτητε οι αλλαγέ, οι οποίες ακόμα και αν ήταν κακές έπρεπε να γίνουν. Λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα των αλλαγών και όχι μόνο τα μειονεκτήματα αυτών που δεν αλλάζουμε. Αυτό είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ο Πέτερ έχει δίκιο μέχρι τώρα λέει ότι η ισορροπία θα πρέπει να διατηρηθεί και ότι οι επιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη των νέων προτάσεων και μέτρων. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την πίεσή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πολίτης επηρεάζεται από τα μέτρα που παίρνει η Επιτροπή και έτσι η Επιτροπή πρέπει να επηρεαστεί και από εμά. Κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι κ. Κάμφρεν έθεσε ένα ερώτημα και προς την Κομισιόν. Με την άδεια του εισηγητή θα ζητήσω λοιπόν από την Επιτροπή να πάρει το λόγο. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσετε την ε, θέση του Κοινοβουλίου στο χρονοδιάγραμμά σας. Θα ήθελα και εγώ να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν, εάν θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Αλμούνια έχει τονίσει πόσο σημαντικό βρίσκει το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους άλλους εμπλεκομένους και τα κράτη-μέλη. Θέλει να κάνει την ε, αναθεώρηση αυτή με πλήρη διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπον τώρα το χρονοδιάγραμμα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ασύμβατο εμείς περιμένουμε ακόμα τα σχόλια από τους εμπλεκομένους και από τα κράτη-μέλη. Θα συνεχίσει η συζήτηση μέχρι το τέλος του μηνός και μετά τον Νοέμβριο θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Ενδιαμέσως συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σας και με άλλους εμπλεκομένους και θα πάρουμε υπόψη όλα τα σχόλια τα οποία διατυπώθηκαν σήμερα και που σίγουρα θα διατυπωθούν και τις επόμενες ημέρες και μήνες και ελπίζουμε ότι αν το Νοέμβριο έχουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου, μπορεί ακόμα να ληφθεί υπόψη. Ο Επίτροπός μας είπε ότι θα ε, ήθελε να έχει το νέο κείμενο για να εγκριθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν όλα πάνε προς ευχήν, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου μπορεί να γίνει η έγκριση του κειμένου αυτού, οπότε μπορούμε να λάβουμε υπόψη όλα τα σχόλια που θα πάρουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και επανέρχομαι στον εισηγητή τον κύριο Ζήμων. Ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική αυτή συζήτηση. Ε, θα ήθελα ως απάντηση σε μια ερώτηση που έκαναν πολλοί συνάδελφοι για την ε, πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μεταχείριση θα τις επιφυλάξουν. Αυτό είναι θέμα πραγματικά κρίσιμο και κομβικό. Εδώ υπάρχει το εξής δίλημα. Είτε θα το εξαιρέσουμε τελείως και θα πούμε ότι έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμβιβαστική διαδικασία για να προσθέσουμε στοιχεία στην πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δώσουμε τη δική μας γνωμοδότηση. Τελείως ελεύθερη πάσης ιδεολογίας. Βλέπουμε, λαμβάνουμε όλη γνώση των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουμε και θέση τώρα εκτός από γνώση ε, όχι το άρθρο 14 ε, προ, ε, το πλαίσιο που προτείνει ναι, όχι, προς Θεού, ποτέ, να αποφύγουμε τέτοιες δηλώσεις. Ο Επίτροπος Αλμούνια ήδη από το καλοκαίρι που είχα την ευκαιρία να του συναντήσω, έχω την αίσθηση ότι έχει την ίδια αντίληψη. Είναι ε, πρόθυμος να συμπεριλάβει και αυτά που θα πούμε. Βέβαια δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά το γεγονός ότι έχουμε έρθει σε αυτή τη δινή κατάσταση σήμερα δεν φταίει η Κομισιόν, γι' αυτό φταίει το Κοινοβούλιο. Καμιά φορά ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει τις προτάσεις της, μα την πρώτη πρόταση την έφερε το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μας εμπόδιζε τίποτα να αρχίσουμε τις εργασίες από το Μάρτιο. Εγώ Είχα ακριβώς πέντε μήνες για να γράψω μια έκθεση. Δεν θα πρέπει να το προσάπτουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την κατηγορούμε που έχει τώρα χρονικό πρόβλημα και πίεση να φέρει την αρρύθμιση. Ίσα ίσα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο Αλμούνια και τους υπαλλήλου ε, για το επικοδομητικό τους πνεύμα και τη στάση τους γενικά στη συνεργασία. Λοιπόν, ποιες είναι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ κυρία Εσαΐα ότι το θέμα της κατανόησης, της συνεννόησης, εάν ε, το καταλαβαίνουν αυτό οι δήμοι κοινότητες, αν τους βοηθούμε για την απόφαση Altman, την είπα. Όποιος δεν καταλαβαίνει την εξήγηση για τα τρία πρώτα κριτήρια, ε, τι να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε, ούτε έχει καμιά θέση ως εμπορικός ε, φορέα στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και με αυτά που είπε ο κύριο Κανφέ και η κυρία Ινετφέλτ, αλλά και εσεί κυρία Σαΐα. Στα πλαίσια των συμβαστικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να κοιτάξουμε και να συζητήσουμε συγκεκριμένα τους κανόνες de minimis. Να ασχοληθούμε με την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής συγκεκριμένα. Ιδιαίτερα το μέγεθος των Δήμων και Κοινοτήτων ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα και υπό την έννοια της συνεργασίας των Δήμων και Κοινοτήτων ή μεγαλύτερους Δήμους που έχουν προβλήματα σίγουρα θα ε, μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση και η πρόταση κυρίας Οκονή το ανέφερα προηγουμένως. Χαίρομαι που η αρχή της επικουρικότητας γίνεται δεκτή και τονίζεται και από όλους τους συναδέλφους και στις τροπολογίες τους. Και βεβαίως συμφωνώ με την άποψη ότι και δυστυχώς έφυγε ο κύριος Χιόκμα, ότι η επικουρικότητα δεν θα πρέπει να είναι πρόφαση για να διατηρηθούν ε, εν λειτουργία προβληματικές εταιρείε. Έχω όμως να πω το εξής και μάλιστα ξεκάθαρα. Μπορεί κανείς να επιθυμεί την απόδοση και το κοινοβούλιο να προσπαθεί να την πρόθει, αλλά σας παρακαλώ να περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί νομική βάση, γιατί το δίκαιο ανταγωνισμού δεν τη δίνει νομική βάση, να ορίζει κάποιου κανόνε, τότε ε, πραγματικά αυτό είναι προηγούμενο και ε, υπερβαίνει τα εσκαμένα. Θα πρέπει με συμπερίληψη του Κοινοβουλίου να προχωρήσουμε σε μια κανονική νομοθετική διαδικασία και όχι στα πλαίσια μιας νομοδότησης που τώρα θα έρθουμε να δώσουμε, αλλά μια απόφαση που στο τέλο, θα διαμορφώσει πώς θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε για την αποδοτικότητα, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει αυτό. Σημείο δεύτερο, σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα και τη μη διατήρηση προβληματικών εταιριών. Συμφωνώ και ευγνωμονώ τον συνάδελφο Σκίνερ που και εδώ έκανε αυτή τη συζήτηση χωρίς ιδεολογία. Κανείς δεν θέλει να συντηρεί προβληματικές επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν. Ο καθένας έχει την άποψη του συναδέλφου Χέρκμαρκ ότι θέλουμε και πρέπει να υποστηρίζουμε τους πολίτες και όχι τις επιχειρήσεις. Μα ακριβώς σκεπτόμενοι τον πολίτη θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάποια στρεβλά και κακό του παρελθόντος. Θα ανέφερε ο κύριος Σκίνερ και ο κύριος Χιόκμαν είπε το θετικό της τηλεπικοινωνίας. Και σε αυτό το τομέα μπορούμε να δούμε κάποιες τρευλές εξελίξεις. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να βγάλουμε και τα διδάγματά μας από το παρελθόν. Αρκεί να σας πω το εξής, ευρυζωνικότητα. Όταν οι τηλεπικοινωνίες ήταν ακόμα θέμα δημοσίου συμφέροντος, ακούσαμε ποτέ ε, ότι θα πρέπει και στην τελευταία ε, ε, γωνιά κάθε χώρας να φτάσει η ευρυζωνικότητα και να την πληρώνει το δημόσιο. Πέρα από όλα τα πλεονεκτήματα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι σήμερα δεν είμαστε πια στην ίδια κατάσταση. Έχουμε ένα νέο κόσμο τηλεπικοινωνιών και χαιρόμαστε που δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες και φροντίζουν να φέρουν ευρυζωνικότητα σε πολλά σημεία των χωρών μας που σίγουρα στο παρελθόν δεν θα ε, είχαμε ή δεν θα είχαμε σήμερα αν συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση που ίσχυε στο παρελθόν. Λοιπόν, παρακαλώ, χωρίς ιδεολογία, ναι, έχουμε τη δυνατότητα τώρα μέχρι τον Νοέμβριο να κάνουμε προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαπραγματεύσεις ε, και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις προτάσεις μας που θα έρθουν μέχρι τότε, επικοδομητικά, στοχευμένα, ελπίζω και είμαι βέβαιος ως Κοινοβούλιο ότι θα φέρουμε μια καλή πρόταση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Εντάξει, λέει και η πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. 17 Οκτώβριο προβλέπουμε να ψηφίσουμε η Ολομέλεια τον Νοέμβριο ώστε να υπάρξει επαρκώς χρόνος για την Κομισιόν να λάβει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου υπόψη της. Ξαναγυρίζουμε στο σημείο της σημείωσης διάταξης παριθμών 6 που αναβλήθηκε χθε. Μία νέα στατική για την πολιτική καταναλωτών και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον Αλφρέντο Παλόνε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Χθες ήμουν αδιάθετος και δεν μπόρεσα να έλθω εδώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν για τις τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν από τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες αυτές συνιστούν τη θέμενη αξία στην έκθεσή μου. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα σας στείλω το τελικό κείμενο λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας. Να περάσω ίσως σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την τροπολογία 1, η οποία παρουσιάστηκε από τη συνάδελφα Φάνα. Η κρίση λέγεται ότι χτύπησε κυρίως τις ε, ασθενέστερες οικονομικές τάξεις και θα έλεγα τη, τα χρέη τους. Πράγματι η κρίση χτύπησε ειδικότερα κάποιες κοινωνικές τάξεις ή κοινωνικές κατηγορίες, να το πω καλύτερα. Στην Ιταλία σαν παράδειγμα, ή όχι μόνο στη δική μου χώρα, έχουμε να κάνουμε με μια κρίση η οποία πληρώνεται από τη μεσαία τάξη αν θέλετε, η οποία πιέζεται ιδιαίτερα. Και λέγεται στην τροπολογία ότι η αιτία της κρίσης είναι η υπερχρέωση. Εγώ το βλέπω και ανάποδα. Ε, πράγματι η υπερχρέωση είναι αιτία της κρίσης και πράγματι πολλές οικογένειες δεν καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση στην πίστοση. Η δεύτερη τροπολογία την οποία συμμερίζομαι αναφέρεται στο περιβάλλον και στην αηφορία του περιβάλλοντος. Δεν μπορώ εγώ να συνδέσω την αηφορία του περιβάλλοντος και την έκθεση η οποία αναφέρεται ε, για τα θέματα των καταναλωτών. Και γι' αυτό θα ήθελα εγώ να διαφωνήσω, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, αλλά είμαι έτοιμος να συζητήσω εφόσον υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση μέσω μιας προφορικής τροπολογίας ίσως. Βλέπω εδώ ότι ίσως είναι συνάδελφος Τρεμόζα, όχι, για την 7 θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία για να, για να μην υπάρχουν ε, παρεξηγήσεις. Λέγεται ότι θα πρέπει να έχουν στη γλώσσα τους οι καταναλωτές ε, τις, ε, τα στοιχεία ενημέρωσης. Και δεν διευκρινίζεται αν μιλάμε για την εθνική γλώσσα ή την περιφερειακή γλώσσα εφόσον γίνεται αποδεκτή ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει συμβιβαστική λύση εδώ. Υπάρχει η εννέα πάντα της συναδέλφου Αλφάνα και λέγεται ότι χιλιάδες ε, καταναλωτές έχασαν εκατομμύρια εκατομμυρίων λόγω των κακών συμβουλών τις οποίες ε, είχαν πάρει δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρξει μια καλύτερη ρύθμιση των αγορών αυτών, των οποίων η εποπτεία πριν από την κρίση ήταν ανεπαρκεστάτη. Και γι' αυτό θα ήθελα να βγάλουμε εμείς την αναφορά στις κακές γνώμες ή να πούμε ότι οι κακές γνώμες, συμβουλές είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι η κρίση αυτή που είναι συστημική κατά τα άλλα προκλήθηκε από τις κακές συμβουλές που δόθηκαν στον καταναλωτή. Νομίζω ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι μία από τις αιτίε, αλλά δεν είναι η βασική. Θα ήθελα να το συζητήσω λοιπόν με τους συναδέλφους να να μιλήσουμε και για τις ε, συλλογικές ε, αιτήσει αποζημίωσης, μαζικές ή συλλογικές αιτήσει αποζημίωσης. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση σοβαρή. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση εδώ, αλλά δεν μπορούμε εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση των συλλογικών, εν πάση περιπτώσει προσφυγών, να καταλήξουμε σε αποτελέσματα στα οποία να συμφωνήσει όλο το Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία ε, και για την 10 και για την 11 να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή διατύπωση γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ευαίσθητο το πρόβλημα αυτό. Η σημερινή συζήτηση θεωρώ ότι μπορεί να μας βοηθήσει που βρίσκομαι, να, καταλάβει κανείς που βρίσκομαι και ε, να προκαλέσει και άλλες προτάσεις από πλευράς των συναδέλφων. Μέχρι αύριο το πρωί. Χθες λιποτάκτησα θα έλεγα, αλλά αύριο θα σας στείλω ε, την το τελικό κείμενο. και θα περιλαμβάνει και τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις οι οποίες ε, ε, θα γίνουν ε, απέναντι σε αυτά που λέω και σήμερα. Ευχαριστώ τους κοιόδης συγητές, τους συναδέλφους, τη γραμματεία, ιδιαίτερα τους συναδέλφους που μου απέστειλαν σχόλια, που με βοήθησαν να διατυπώσω σωστά την άποψη και μου έστειλαν τις τροπολογίες τους, τις οποίες όπως είδατε λαμβάνω υπόψη εν πολύ, έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρότασή μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Αντολίν. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πει προηγουμένω ότι ο δεκάλογος που παρουσίασε ο κ. Παλώνη μου φάνηκε πάρα πολύ θετικό, ο δεκάλογος που περιέχεται στην γνωμοδότησή του και θα ήθελα να προσπαθήσω να προσθέσω ορισμένε ιδέε για να συμπληρώσει να συμπληρωθεί αυτό το οποίο λέει ο κ. Παλώνα για τη στρατηγική. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να αυξηθούν, να ανέβουν τα επαγγελματικά πρότυπα, να αποφευθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να υπάρχει και καλύτερη αξιολόγηση κινδύνου από την πλευρά των καταναλωτών. Για τα, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ειδικότητα, είναι σαφές ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτονται από λιγότερη προστασία οι καταναλωτές εκεί από ότι σε άλλες περιπτώσεις. Είναι απαραίτητο επίσης να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή χάρτα καταναλωτών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεν πρόκειται να πω περισσότερο σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικό θέμα. Επίσης, για τη στρατηγική αυτή νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουν και οι εκπρόσωποι των ε, καταναλωτών που βρισκόνται στις ε, εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ε, διευκολύνσει σε τεχνικό επίπεδο και τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνθήκες αντίστοιχε με, αυτόν, με αυτές των εκπροσώπων των βιομηχανιών που φυσικά έχουν αρκετά υλικά μέσα στη διάθεσή τους και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όπως είπε και ο κύριος Παλώνε είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση στις βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και όχι να προσκρούει κανείς σε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν διακριτικό ή αυθαίρετο χαρακτήρα από τις τράπεζες. Περιμένουμε λοιπόν το τελικό κείμενο του κύριου Παλώνε και τις συμβαστικές τροπολογίες και νομίζω ότι είναι πολύ θετική η κατεύθυνση που έχει αναλάβει ο κύριος Παλώνε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Η Σόφη συντομοτάτη θα σταθώ Έχουμε πάρει μια σειρά από συμβαστικές τροπολογίες που πιστεύω ότι μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Έχουμε κάνει δύο προτάσεις για ίσονες τροποποιήσεις. Δεν είχαμε βέβαια την ευκαιρία να συζητήσουμε ακόμα με τον κύριο Παλώνε, αλλά νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ βρισκόμαστε στη συμφωνία και υποστηρίζουμε την πρόταση του κύριου Παλώνε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση. Αλφρέντο, θες να ξαναλάβεις το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα όπως συνηθίζουμε. Επαναλαμβάνω <clears throat> ότι θα περιμένω τους συναδέλφους μέχρι αύριο το πρωί να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Πραγματικά γνωρίζουν οι συναδέλφοι ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο όχι μόνο στον τομέα της ενημέρωσης αλλά και στον τομέα της κατάρτισης. Θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις δύο θέσεις γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι μόνο με τεχνικούς στόχους και λεπτομέρειες τεχνικές δεν θα πετύχουμε. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να στογεύσουμε καλύτερα αυτόν τον συσχετισμό στον οποίο προαναφέρθηκα, όλοι από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει στην 11η Οκτωβρίου η τελική ψηφοφορία 17 και κανονικά θα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια, την πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Νομίζω ότι κλείσαμε για σήμερα το πρωί. Στις 3 η ώρα ξέρετε ότι έχουμε τον νομισματικό διάλογο με τον Ζαν